Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to this afternoon session of the Internal Market Committee. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σήμερα το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών θα ξέρετε ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου έφερε σε εμά το θέμα αυτό, αλλά εννοείται ότι θα συνεργαστούμε και με την Οικονομική Επιτροπή. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε την εξή διαδικασία, να προσκαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει τη δικιά τους έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς σκέφτονται να εξετάσουν και να αναλύσουν το θέμα αυτό με μια έκθεση αντικτύπου. Είναι θέμα λοιπόν τραπεζικών λογαριασμών, πώς μπορεί κανείς να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό χωρίς εμπόδια, γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο για τους πολίτες να ανοίξουν, τους φαίνεται πολύ πολύπλοκο ή δεν ξέρουν τις διαδικασίες πώς πρέπει να το κάνουν, πώς να ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Είναι λοιπόν σωτική σημασία για τους πολίτες αυτό το θέμα και εμείς μπορούμε να το εξετάσουμε. Οπότε θα στήσω από τον κύριο Φιλίπ Πελέ που είναι επικεφαλής ε, της σχετικής μονάδας στην Επιτροπή να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό με διαφάνειες. Και στη συνέχεια ζητήσαμε από την κυρία Γκέμπαρτ που είναι η συγγήτρια να έρθει εδώ και ο Hans Peter Μάιρ που είναι σκιώδης, Ashley Fox, Σμιτ δεν έχουν έρθει ακόμα. De Jong, ούτε αυτός έχει έρθει ακόμα, Σαλβίνη και οποιοδήποτε άλλο σε θέλει το λόγο. Έχουμε χρόνο λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα χωρίς άλλη καθυστέρηση εκτός αν η κυρία Γκέπερ θέλει εισαγωγικά να κάνει κάποια σχόλια ή μια και καλή μετά την παρουσίαση. Τι προτιμάτε. Έχετε κάτι να πείτε εισαγωγικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Όπως ε, είπες και εσύ, είναι όντως ε, πολύ σημαντικό το θέμα που συζητούμε σήμερα και σήμερα ακριβώς με σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε, η πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί αλλιώς δεν μπορεί κανείς να, να λειτουργήσει ως άνθρωπος, γιατί ε, κάποιος δεν μπορεί να μην θεωρείται ουσιαστικά άνθρωπος αν δεν έχει ε, τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε η πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω πολλών τρόπων, γιατί εδώ δεν μιλούμε μόνο για ανθρώπους που ε, εισπράττουν πολύ λίγα, λίγα χρήματα. Μιλούμε επίσης και για άτομα που έχουν δικαίωμα να μην την χάνουν διακριτική μεταχείρισης όπω βεβαίω όλοι. Ε, έχουμε και το φόρουμ της Κρακοβίας ε, προχτές, το οποίο συζήτησε επίσης ένα, ένα τέτοιο, το, ίδιο ακριβώ ζήτημα και υπήρξε ένα παράδειγμα όπου μια γυναίκα νέα πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό θέλει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα και της λένε ναι μπορείτε να νοικιάσετε το διαμέρισμα εάν μας δώσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό πηγαίνει στην τράπεζα και της λέει «Α, η τράπεζα λυπούμε, όταν δεν έχει, α, εφόσον δεν έχετε έδρα στη χώρα δεν μπορείτε να ανάξετε λογαριασμό». Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το μπρος πίσω είναι ε, προβληματικό και δεν έχει καθόλου πρόσβαση αυτή η γυναίκα τελικά στη χώρα στην οποία θέλει να σπουδάσει. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και από αυτού πρέπει να εργαστούμε κι εμείς. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εδώ και χρόνια ζητούμε να υπάρξει πρόσβαση, να ανοίξει η πρόσβαση. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ επίσης μας υποσχέθηκε στα πλαίσια των συζητήσεων για την πράξη για την εσωτερική αγορά ότι αυτή θα αποτελέσει μία από τις προτεραιότητές του. Τώρα έχουμε αυτές τις προτάσεις τις οποίες υποβάλλει η Κομισιόν. Ειλικρινά έχω απογοητευτεί. Απογοητεύτηκα γιατί εδώ μιλούμε απλώς για απλές συστάσεις. Δεν είναι τελικά οδηγία, δεν είναι σχέδιο οδηγίας αυτό που υπέβαλε η Κομισιόν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε κι άλλο με την Κομισιόν. Η ανακοίνωση ή απλώ μια σύσταση προ τα κράτη-μέλη ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Εντάξει, καλή είναι, αλλά ξέρουμε πώ τελειώνει το πράγμα, που, καταλήγει. Δεν γίνεται τίποτα και αυτές οι δυσκολίες που υπάρχουν προφανώς συνεχίζονται γιατί το ε, εξακολουθεί να ισχύει το, δίκαιο, το ε, δίκαιο συγγνώμη, το εθνικό του κρατου μέλους. Οι συστάσεις απλές συστάσεις είναι, δεν μπορούν να υποχρεώσουν το κράτος μέλο να αλλάξει το δίκαιό του. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να συζητήσουμε είναι κάτω από ποιε προποθέσει θα επιτρέψουμε αυτό το δικαίωμα σε πρόσβαση σε τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί υπάρχουν και τα συμφέροντα της ε, τράπεζας προφανώς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι τράπεζες μπορεί να έχουν ε, να, κάποια ανησυχία για το ότι μπορεί να χάσουν χρήματα. Ε, υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Και επίσης πώς ε, τι θα πρέπει να, πώς θα πρέπει να είναι μια κάρτα τραπεζική, ποια δικαιώματα θα πρέπει να δίνει στον κάτοχό της. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ερωτήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία πρέπει να απαντηθούν για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Όπως είπα στην αρχή είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους τους πολίτες σε αυτόν τον πολύ υψηλή τεχνολογία και γρήγορο κόσμο που ζούμε, να δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται και νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι ένα ε, γενικό ε, δικαίωμα που έχουν οι πολίτε να έχουν πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να μπορούν να υποφελούνται από τις υπηρεσίε, οι οποίε επίση συνδέονται με την ύπαρξη αυτού του λογαριασμού. Ευχαριστώ. Good. Thank you for that very... Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την καλή εισαγωγή. Ας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας παρουσιάσει την έκθεση αντικτύπου που έχουν κάνει και τις συστάσεις τους για το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο κύριε Πελέ, έχουμε τις διαφάνειές σας, τις βλέπουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Γκέπαρτ και όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές εδώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την έκθεση αντικτύπου που συνοδεύουν βέβαια τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πρόσβαση σε ε, τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών. Πρώτα απ' όλα, πώς έχει το πρόβλημα. Ποιο είναι το πλαίσιο. Όπως είπε και η κυρία Κέπαρτ, πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι κάτι στοιχειώδες προκειμένου να μπορεί κανείς να συμμετέχει στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Για σκεφτείτε το, χωρίς λογαριασμό τραπεζικό, τι θα μπορούσατε να κάνετε. Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι θα μπορούσα να κάνω. Τίποτα. Τι θα κάνω; Κάθε φορά θα πρέπει να πηγαίνω στην τράπεζα για να ε, παίρνω λεφτά. Τώρα έχω συνηθίσει να το κάνω αλλιώ με την κάρτα μου, το μηχάνημα. 30 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λογαριασμό. Η δυσκολία είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς ε, τα 30 εκατομμύρια που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό γιατί δεν θέλουν να τον έχουν ή από την άλλη μεριά έχουμε και εκείνου οι οποίοι θα θέλουν αλλά δεν μπορούν ή δεν τολμάνε να ζητήσουν να τους ανοίξει μια τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό. 30 εκατομμύρια λοιπόν δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Πρόκειται για ανθρώπου συχνά που έχουν ε, χαμηλά ε, έσοδα, αλλά όπως λέει και η κυρία Γκέπαρτ, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν πολλές φορές να μπορούν και να κυκλοφορούν σε διαφορετικές χώρες, που είναι μια από τις στοιχειώδεις ε, ελευθερίες που έχουμε στην Ευρώπη. Αλλά αν πάνε σε μια άλλη χώρα δεν μπορούν να ανοίξουν εκεί εύκολα τραπεζικό λογαριασμό, ούτε οι εποχιακοί που μετακινούνται, ούτε συνταξιούχοι που πάνε αλλού για να περάσουν ε, τη σύνταξή τους ενδεχομένω κλπ. Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και 91% του πληθυσμού, των ενηλίκων δηλαδή της Ευρώπης των 12, ε, ενώ 97% στην Ευρώπη του 15. Ο μέσος όρος της Ευρώπης των 12 ε, Βέβαια, επηρεάζεται και από την περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπου εκεί οι τραπεζικές υπηρεσίες δεν έχουν αναπτυχθεί πολύ. Εκεί είναι λοιπόν πολύ πιο χαμηλό το ποσοστό, 50%. Θεωρούμε πάντως ότι το να μην έχει κανείς ένα τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία δεν είναι τόσο προβληματικό όσο να μην έχει κανείς λογαριασμό στη Γαλλία ή στις Ηνωμένες γιατί κυκλοφορεί πολύ το ρευστό, χρησιμοποιούν πολύ το ρευστό στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ακόμα. Αλλά αλλού όπου ηλεκτρονικές ε, ε, πληρωμές είναι η καθημερινότητα, εκεί ο κόσμος που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα πάντως για την κατάσταση αυτή όχι όσο θα θέλαμε. Πάντω, όταν γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις και ό,τι μελέτες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν ρωτάμε τις τράπεζες, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κόσμο λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και η δίκηση στις χώρες μέλη λέει επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό όμως με το οποίο δεν συμφωνούν είναι το μέγεθος του προβλήματος. Πολλέ χώρε μέλη σε δημόσια διαβούλευση επιμένουν ότι πρέπει να υπάρχει και ελαστικότητα. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει δράση μέχρι τώρα όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το ένα είναι η ζήτηση από τους ίδιους τους καταναλωτές που μπορεί για ψυχολογικούς λόγους ή για άλλους λόγους να μην κάνουν το βήμα να ζητήσουν ένα λογαριασμό, είτε γιατί τους λείπει η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, η αυτοεκτίμηση και δεν πάνε στην τράπεζα να πούνε ανοίξτε μου ένα λογαριασμό. Μπορεί να υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Και έτσι όπως έχει κατάσταση σήμερα, μάλλον θα επιδεινωθεί αυτό το πρόβλημα αντί να βελτιώνεται. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Έπειτα έχει να κάνει και με το θέμα του οικογενειακού προπολογισμού. Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα λένε ότι είναι πιο εύκολο να ελέγξεις τις δαπάνες σου του τι έχει στο πορτοφόλι σου, κοιτώντα μάλλον τι έχει στο πορτοφόλι σου, παρά κοιτώντα ε, το εκαθαριστικό τη τράπεζας που σου στέλνει. Η Επιτροπή πάντως και ο ΣΑ έχουν κάνει κάποιες ε, προσπάθειες για να έχουν περισσότερα δεδομένα. Έπειτα ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, αρκετή πληροφόρηση για να ξέρει ε, κανείς ε, πώς αποφελείται από το άνοιγμα ενός λογαριασμού εφόσον μπορεί να έχει χαμηλό κόστος βέβαια η συντήρηση ενός τέτοιου λογαριασμού. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ένας ε, όντως λόγος για τον οποίο δεν ζητούν ε, τραπεζικό λογαριασμό πολλοί άνθρωποι είναι ότι έχει κάποιο κόστος. Δεν έχει αναπτυχθεί πολύ ο τραπεζικό τομέα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπω είπαμε και πριν, γι' αυτό και ο κόσμο ε, στι συναλλαγέ του χρησιμοποιεί πολύ συχνά ρευστό. Πάντω το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά βασικά προϊόντα, απλά προϊόντα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις απλές ανάγκες που έχουν οι πολίτες αυτοί. Όταν είσαι φοιτητή, δεν χρειάζεσαι hedge funds, δεν χρειάζεσαι δύσκολα πράγματα, έναν απλό λογαριασμό θέλεις. Και επιπλέον, Υπάρχουν και κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις νομικές για να έχεις πρόσβαση σε λογαριασμό. Πρέπει να έχεις μια διεύθυνση στη χώρα στην οποία θες να ανοίξει λογαριασμό για να καταπολεμηθεί βέβαια το ξέπλυμα παράνομου χρήματος. ή άλλες πρακτικές, οι τράπεζες δεν είναι πρόθυμες να ανοίξουν λογαριασμό σε κάποιον ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια, στην επικράτεια γιατί αν φτάσει στο μείον ο λογαριασμός είναι πολύ δύσκολο να πάρει πίσω τα λεφτά της η τράπεζα γιατί το άτομο αυτό μπορεί να έχει φύγει, να έχει πάει στο εξωτερικό και για να καταφέρει να πάρει πίσω τα λεφτά της η τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να ξοδέψει στην προσπάθεια αυτή. Και ένας άλλος λόγος είναι το θέμα του κέρδους. Η τράπεζα δεν θέλει, δεν είναι πολύ πρόθυμη να ανοίξει λογαριασμό σε κάποιον που έχει χαμηλά εισοδήματα γιατί φοβάται ότι δεν θα έχει αρκετό κέρδος από τις καταθέσεις του. Υπάρχει όμως και μια συμμετρία πληροφόρησης. Οι τράπεζες προτιμάνε να μιλάνε και να ενημερώνουν τον κόσμο που έχει περισσότερα χρήματα παρά αυτούς που είναι χαμηλών εισοδημάτων. Μπορεί να ετοιμάζει έτσι, για μπροσούρες, οι οποίες καταλήγουν βέβαια στα χέρια εκείνων που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, αποκλείοντας συγχρόνως τους ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων. Όπως θα έπρεπε οι τράπεζες να έχουν το θάρρος να δώσουν σημασία και στα χαμηλά εισοδήματα. Και κάποιες τράπεζες, μια ισπανική για παράδειγμα που δραστηριοποιείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέληξε στο ότι μπορεί να κάνει κερδοφόρες business σε συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς χαμηλών εισοδημάτων. Οπότε σιγά σιγά άρχισε να τους προσφέρει πρώτα τον βασικό λογαριασμό πληρωμών και σιγά σιγά άρχισε να τους προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες ήταν κερδοφόρες για την τράπεζα τελικά. Ποιε είναι οι συνέπειε τώρα για του καταναλωτέ πρώτα απ' όλα, άμα δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα, αν δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ δύσκολο να αγοράσει το οτιδήποτε από το διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει τι διευκολυνσει που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία η οποία προσφέρει υπηρεσίες. Ας πούμε μπορεί να εκμεταλλευτεί εκτόσεις που κάνει μια επιχείρηση στις πωλήσει της μέσω διαδικτύου. Βέβαια κοστίζουν και αυτές οι συναλλαγές και ας ακούγεται περίεργο. Είναι όμως αλήθεια. Έπειτα στιγματίζεται το κομμάτι αυτού του πληθυσμού που δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό. Έπειτα αναφερθήκαμε πριν και στην μετακίνηση των ανθρώπων από χώρα σε χώρα. Όντω αποτελεί εμπόδιο. Ε, είσαι φοιτητή, Θε να πας αλλού να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίε. Δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό εκεί. Αυτό δεν αμαυρώνει την εικόνα της Ευρώπης. στην ε, Ευρώπη δεν έχουμε σύνορα, μπορούμε να μετακινηθούμε, το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Έπειτα, ο κλάδος, όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά γενικότερα είναι μια χαμένη ευκαιρία. Σας είπα, τράπεζες έχουν βρει τρόπο να έχουν ε, συναλλαγές με τα άτομα χαμηλών εσόδων, αλλά και άλλοι που πουλούν μέσω διαδικτύου αυτοί δεν ε, έχουν σαν πελάτες τα άτομα που δεν έχουν ε, τραπεζικό λογαριασμό. Ε, φοβούνται οι άνθρωποι ότι όταν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους μέσω διαδικτύου έχουν να πληρώσουν κάτι παραπάνω, ενώ ρευστό δεν χρειάζεται. Όμως αν πρέπει να πληρώνουν ρευστό σημαίνει ότι όλες αυτές οι εταιρείε είτε είναι ηλεκτρισμού είτε είναι οτιδήποτε θα πρέπει να έχουν ένα γραφείο όπου να έχει πρόσβαση ο κόσμος για να πληρώνει σε ρευστό. Αυτό τους κοστίζει όμως των επιχειρήσεων αυτών και δεν το θέλουμε. Στον Ηνωμένο Βασίλειο ίσως να ξέρετε ότι ο κλάδος ήθελε να δημιουργηθεί ε, αυτό, δηλαδή να είναι υποχρεωτικό το να έχει τραπεζικό λογαριασμό ο καθένας και το θέλω αυτό και το κράτος γιατί έτσι θα κόστιζε λιγότερο η επίδοση των συντάξεων. Άρα λοιπόν ο στόχος μας επ' αυτού, για να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, οι στόχοι μας. Ε, μίλησα για τα άτομα χαμηλών εισοδημάτων, αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτούς. Πρόκειται για διάφορους ενδυνάμει πελάτες που είναι σε κανονική εντό εισαγωγικών κατάσταση. Γι' αυτό και προτείνουμε, μάλλον συστήνουμε, πλήρη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Διασφαλίζοντας προσφορά υπηρεσιών πληρωμών από τις τράπεζες με προϋποθέσεις που να είναι ικανοποιητικέ για όλου. Έτσι ώστε οποιοδήποτε δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό να μπορεί να το κάνει και να μην εμποδίζεται από την οικονομική του κατάσταση. Στόχοι μας είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως πρέπει να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλά ακούμε για τη σύσταση αυτό. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση. Χρειάζεται, επειδή οι περισσότερες χώρες δεν έχουν εξετάσει το θέμα αυτό σε εθνικό επίπεδο. Και αυτές που το έχουν κάνει, σε 11, Το έκαναν για διαφορετικούς λόγους. Η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν νομοθετήσει σχετικά το Ηνωμένο Βασίλειο, οι χώρε. Ζήτησαν από το κλάδο να εκπονήσει έναν κώδικα δεντολογίας και να φροντίσει για την πρόσβαση. Η Γερμανία επίσης. Ξέρουμε ότι εκεί όπου υπάρχει αυτός ο κώδικας, πριν από χρόνο πριν από ένα χρόνο συζήτησαν και το ενδεχόμενο νομοθεσία. Στι κάτω χώρε γίνονται και συζητήσει στο Κοινοβούλιο από αυτού. Στη Δανία, τη Σουηδία και σκανδιναβικέ χώρε υπάρχουν γενικέ αρχέ. αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες ούτε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εκτός από την Φιλανδία πάντως δεν υπάρχει πλαίσιο για τη διασυνοριακή πρόσβαση. Θεωρούμε ότι δεν λειτουργεί συνεπώς αρκετά ικανοποιητικά η εσωτερική αγορά σε αυτό το τομέα και ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Αν δεν κάνουμε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Αν δεν υπάρξει κάποιο πολιτικό μήνυμα δεν θα γίνει τίποτα. Οι τράπεζες έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν αυτή την εποχή. Ούτε οι εθνικές αγορές μπορούν να βοηθήσουν αν δεν υπάρξει κάποια όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν δισταγμοί από την τραπεζική βιομηχανία και αυτό είναι κατανοητό γιατί τέτοια μέτρα που δίδουν εγγυήσεις πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες πιστοτικές Όπως είπα, ε, τα δεδομένα δεν είναι ε, πάρα, πολλά που έχουμε στη διάθεσή μας και πολλά αμφισβητούνται. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να αξιολογήσουμε μια πρόταση. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή θα είναι λειτουργική και θα καλύπτει μέρος του προβλήματος. Τώρα για το επίπεδο της τιμής του τραπεζικού λογαριασμού και αν θα πληρώνεται από τους καταναλωτές ή όχι. Οι τράπεζες ε, θα πρέπει να υποστηρίξουν ότι δεν χάνουν χρήματα από τη διαδικασία αυτή και αν χάνουν χρήματα τότε θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός για να αντισταθμίσει τις απώλειές τους. Βλέπετε εδώ μια υψηλή υπόθεση, ένα υψηλό σενάριο, ένα χαμηλό σενάριο και ένα μέσο ουδέτερο το κόστος, το μέσο κόστος, το οποίο είναι 55 ευρώ, τότε έχουμε μια καθαρή δυνατότητα κέρδους 3 ευρώ για τον παροχέα της υπηρεσίας και γενικά όλες οι κατηγορίες ε, μπορεί να κερδίσουν αλλιώς ευθυνότερο, σε ευθυνότερη κοστολόγηση του λογαριασμού, τότε η βιομηχανία, η τραπεζική ίσως να μην κερδίζει, αλλά να χάνει αντίθετα κάποια ποσά. Αν λοιπόν σε 13 ευρώ, ευρώ συγγνώμη, παίρνουμε τη βελγική εμπειρία, όπου ένας βασικός λογαριασμός κοστίζει ακριβώς 13 ευρώ το χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση και αν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, η τραπεζική βιομηχανία θα πρέπει να πληρώσει ένα κόστος συνολικά 400 με 500 εκατομμύρια. Αλλά οι καταναλωτές θα κερδίσουν, θα εξοικονομήσουν τέσσερις φορές το ποσό αυτό. Και στα κράτη-μέλη αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει αντιστάθμιση αποζημίωση των τραπεζών από τα κράτη. Λόγω όλων αυτών λοιπόν προτείνουμε ένα μέσο το οποίο συνιστά ουσιαστικά μια σύσταση και μια πολιτική επιλογή. Η σύσταση είναι το πιο ευέλικτο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε ένα ξεκάθαρο και έγκαιρο μήνυμα στα κράτη-μέλη στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που οργανώσαμε το 9 και το 10 από τις διαβουλεύσεις αυτές βγαίνει ότι σίγουρα η σύσταση δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η οδηγία αλλά όπως είπε ο αρμόδιος επίτροπος τον μήνα Ιούλιο όταν έγινε δεκτή η σύσταξη, η σύσταση, συγγνώμη. the Commission uh, will consider a possibility of legislating. Και πριν κλείσουμε, αυτό το οποίο προτείνουμε στα πλαίσια της σύστασης είναι ένα απλό προϊόν, έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να καταθέτει, να αποσύρει, θα συνοδεύεται από μια ηλεκτρονική κάρτα, γιατί είναι κάτι το απαραίτητο στην κοινωνία μας σήμερα. Δεν προβλέπουμε όμως κάποια δυνατότητα υπερανάληψης. About issue of, of debt recovery with people that may run the Λοιπόν, κάποιος που θέλει να χρησιμοποιήσει την κάρτα του για να αποσύρει περισσότερα από όσα έχει στο λογαριασμό, τότε θα υπάρχει, θα προβλέπεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Και αν δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη, τότε η συναλλαγή δεν θα ολοκληρωθεί. Θα εμποδιστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμποδίζει, αλλά και προστατεύει τον καταναλωτή από υπερχρέωση ή θα προκαλέσει υπερβολικό κόστος. Για τις συνθήκες πρόσβασης αναφέρθηκα, ο λογαριασμός αυτός θα είναι ανοιχτός σε, όλον σε όλους τους καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κάτι τέτοιο, για να διευκολύνουμε και την εσωτερική πρόσβαση, όπως επίσης και την ε, διασυνοριακή. Η τιμολόγηση. Προφανώς εδώ υπάρχει ένα θέμα για το κόστος της ε, βιομηχανίας της πιστοτικής. Οι λογαριασμοί αυτοί θεωρούμε ότι είτε θα είναι δωρεάν γιατί ισχύει σε διάφορα κράτη-μέλη και γιατί να αλλάξει άραγε. Ή με μια ελάχιστη τιμή κόστους για τον καταναλωτή. Ε, θα πρέπει φυσικά τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για το επίπεδο τιμολόγησης του λογαριασμού. Λοιπόν, θεωρούμε ότι έχουμε ένα πολύ ευέλικτο μέσο στη διάθεσή μας, είναι ένα μέσο το οποίο στέλνει το σωστό μήνυμα και τώρα θα πρέπει σε εννέα μήνες να δούμε αν το μήνυμα ακούστηκε, αν τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δράση για να εφαρμόσουν όχι τις συνταγές αλλά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ για μια συνοπτική και χρήσιμη ανάλυση Έχουμε αρκετά από τα έγγραφα στα οποία αναφερθήκατε εδώ μαζί μας. Καλώς. Η συγγήτρια μας είναι η κυρία Γκέπχαρτ. Έχουμε επίσης και τον κύριο Μάιερ. Και ο Σμίτ είναι απόν συνεισηγητής. Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι εδώ. Και του τους πράσινους κάποιος δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, να ακούσουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Η κυρία Γκέπχαρτ ήδη μίλησε. Θέλετε να ξεκινήσετε ή στο τέλος. Τι προτιμάτε. Λοιπόν, να ακούσουμε τους κοιόδης πρώτα. Ο κύριος Μάγερ, Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν ε, για όλα όσα μας παρουσίασε και που έχει κάνει και όλη την ε, εργασία που πρέπει. Αυτή η αξιολόγηση κόστους και ωφέλειας ε, δεν κατάλαβα πώς ακριβώς έχει ενσωματωθεί στο κείμενο. Μήπως μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα παραπάνω. Συνολικά νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι πεπισμένο ότι όντως υπάρχουν πολύ περισσότεροι που χρειάζονται ε, ε, να έχουν ε, λογαριασμό, αλλά οι περισσότεροι τον έχουν είτε επειδή τους τον έχουν ανοίξει οι γονείς τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αλλά έναν βασικό, ένα βασικό λογαριασμό τον χρειάζονται όλοι. νομίζω λοιπόν ότι ένας απλός λογαριασμός είναι αυτό που χρειάζεται. Και ίσως να πρέπει να το πούμε πιο παραστατικά στο κείμενο, δεν μιλούμε για δάνεια, δεν μιλούμε για υπεραναλήψεις κτλ. Μιλούμε για έναν απλό λογαριασμό. Επίσης, όπως και η συγγήτρια, και εγώ είμαι της άποψης ότι η σύσταση δεν αρκεί. Έχουμε θέσει πολλά ερωτήματα, έχουμε συζητήσει πολύ στα κράτη-μέλη και στη Γερμανία επίσης, γιατί επισήμως λένε τα κράτη-μέλη ότι μα, το σύστημα λειτουργεί για μας, οι τράπεζες μας είπαν ότι δεν υπάρχει καμία ε, άρνηση, ή, ε, ε, ε, όταν κάποιος ζητάει να ανοίξει λογαριασμό τον ανοίγει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κτλ. Αλλά τελικά το, το σύστημα δεν δουλεύει τόσο καλά όσο θέλουν να το παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις ε, συστάσεις και να κάνουμε τελικά να ακούσουμε μια νομική πρόταση από την Κομισιόν. Ε, γιατί η Κομισιόν είπε ότι έχει μιλάει για 30 ε, εκατομμύρια, άτομα ε, τα οποία θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό. μάλλον με μία απλή σύσταση δεν θα τα καταφέρουν να ανοίξουν λογαριασμό αυτά τα 30 εκατομμύρια ανθρώπων. Τέτοια θέματα λοιπόν που πλήττουν άμεσα τους καταναλωτές χρειαζόμαστε σαφής, σαφή κατεύθυνση. Τώρα, στο κεφάλαιο 4 είναι σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Μιλάτε για 55 ευρώ ανά έτος ή για 13 ευρώ το έτος. Ε, εντάξει, είναι λίγο μεγαλύτερο το φάσμα μεταξύ 0 μηδενικού ε, ευρώ ανά έτος ή 200 ευρώ το χρόνο. Ε, υπάρχει και μεγαλύτερη ψαλίδα όπως βλέπετε. Εγώ δεν θέλω να καθορίζουμε αριθμούς, δεν είμαι τόσο υπέρ των συγκεκριμένων αριθμών, αλλά η εσωτερική ε, ε, αγορά έτσι όπως είναι σημαίνει ότι υπάρχει ένα τέλος εντός του, εντός του κράτους, κρατικό τέλος. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο σε πιο ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην παραμείνουμε στα στενά κρατικά όρια. Είπαμε λοιπόν ότι η πρόταση γίνεται στα ε, εν είδη σύστασης, Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εποπτεία των ε, υπηρεσιών των χρηματοπιστωτικών. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ γραφειοκρατική η λύση που ε, έχουμε επιλέξει. Ας έχουμε ένα λογαριασμό απλό, να μπορεί να ανοίξει ο, ο οποιοδήποτε πολίτης ένα λογαριασμό, χωρίς να βλέπουμε τώρα σε πολλές γραφειοκρατίες κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι για το θέμα αυτό θα πρέπει να ρωτηθούμε. Είναι στο συμφέρον του πολίτη, του καταναλωτή να κάνουμε μια σύσταση που κατά την άποψή μου σίγουρα δεν πρόκειται να πάει πουθενά παραπέρα και θα παραμείνει ω σύσταση. Δεν θα γίνει τίποτε άλλο. Ή μήπω πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να κάνει κάτι πιο σοβαρό. Τέλο. Το είπατε εσεί, Πρόεδρε, αγαπητέ Μάλκομ. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που συνδέονται και τα οποία μάθαμε στο στη Κρακοβία. Όταν κάποιο έχει έναν, ε, έναν λογαριασμό, ε, δεν μπορεί να στείλει έμφασμα σε μια χώρα του εξωτερικό γιατί δεν το κάνει η τράπεζα. Ε, οπότε τι νόημα έχει να τον έχει το λογαριασμό. θα πρέπει να, να μπορέσουμε να συνδέσουμε περισσότερο όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να δίνει ένας λογαριασμό στον καταναλωτή. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Mr. Fox. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Πέλε για την παρουσίασή του εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο η ομάδα μου θα πρέπει να καθίσει και να σκεφτεί πριν καταλήξει συμπεράσματα. Πρέπει να σας πω ότι όταν άκουσα την κυρία Γκέπαρτ στις αρχικές της παρατηρήσεις συμφώνησα μαζί της, γιατί το βρήκα φοβερό να μπορεί κανείς στη σύγχρονη ζωή να προχωρήσει χωρίς να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιώντα μόνο ρευστό. Όμως, να, από κάποιο ποσοστό από τους πολίτες μας το κάνει αυτό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε έναν κώδικα διοντολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες προσφέρουν έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών. Υποθέτω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το κύριο κίνητρο ήταν η εξοικονόμηση από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών και θεώρησε ότι θα μπορούσε να το στολίσει αυτό μιλώντας και για κοινωνική ένταξη κλπ. Το σημείο 6 του κύριου Πέλε που αναφέρεται σε ευρωπαϊκή δράση αυτό με ενδιαφέρει πολύ, αυτή η έκτη διαφάνεια του κύρου Πέλε. Δεν νομίζω ότι αυτό που λέτε στέκει, γιατί οι λόγοι που δίνεται είναι να, ότι δεν λειτουργεί αρκετά καλά η εσωτερική αγορά και ότι άρα υπάρχουν ε, περιτά εμπόδια στην κινητικότητα. Μα υπάρχουν και κάρτες μέσα στις οποίες υπάρχει ένα ποσό και οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλαδή το 7% στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, που προτιμάει το ρευστό, μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο αγοράζοντας μια ε, κάρτα ε, χρεωστική. Λέτε ότι η έλλειψη βασικού λογαριασμού πληρωμών αποτελεί εμπόδιο και για την διασυνοριακή κινητικότητα. Αναρωτιέμαι, είναι σωστό αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι οι περισσότεροι που περνάνε από μια χώρα στην άλλη για να πάνε στη δουλειά τους έχουν και δουλειά και έχουν και τραπεζικό λογαριασμό. Δέχομαι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό θα υπάρχει το οποίο ε, μετακινείται για να ψάξει να βρει δουλειά. Κάποιος δηλαδή που θα πάει σε άλλη χώρα χωρίς να έχει δουλειά, επειδή ψάχνει να βρει δουλειά εκεί, κάθε μέρα ε, μου φαίνεται ότι είναι πολύ λίγοι. Συμφωνώ με την κυρία Κέπχαρτ βέβαια ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά αναρωτιέμαι είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση για να διορθωθεί. Αν αφήσετε το κάθε κράτος μέλος να το χειριστεί, όπως κάναμε με τον κώδικα δεντολογίας μας εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως τελικά διαπιστώσετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος λύθηκε. Επανέρχομαι λοιπόν στο αρχικό μου σχόλιο. Δεν είναι κάτι για το οποίο η ομάδα μου έχει καταλήξει. Εσείς κάνατε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, αλλά είμαι επιφυλακτικός πολύ συχνά και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Εντοπίζουμε ένα πρόβλημα και η απάντησή μας είναι κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που μας είπατε είναι αυτό το κάτι. Και άρα πρέπει να το κάνουμε λέτε. Συχνά όμως καταλήγουμε στο να δαπανάμε περισσότερα χρήματα και να δημιουργούμε άλλα μεγαλύτερα προβλήματα και περισσότερη γραφειοκρατία από ότι το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να διορθώσουμε. Με αυτή λοιπόν την επιφύλαξη τελειώνω πρόεδρο και σας λέω ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φόξ. Γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση για την έκθεση αντικτύπου, για να προβληματιστούμε και να μπορούμε κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Ο κύριος Ντεγιόγκη πρώτα, μετά και ο κύριος Χρόσμα και ποιος άλλος θέλει. Τώρα ο κύριος Ντεγιόγκ πάντως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ακριβώ το αντίθετο από αυτό που είπε ο κύριος ε, Φόξ, γιατί ακριβώς εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι συγκεκριμένο για να βοηθάει τους ανθρώπους να εντάσσονται στην κοινωνία και αυτό το 7% που δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό όντως θα έπρεπε να βοηθηθεί. Δεν κάνουμε πολλά για αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε στο 2011 και πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει τόσος κόσμος ο οποίος ε, δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μήπως εδώ πέρα τίθεται και θέμα ανθρωπίνου δικαιωμάτων. Μήπως έχει το θέμα να κάνει με τις εξελίξεις της κοινωνίας μας. Τώρα, δώσατε τα επιχειρήματά σας και είπατε γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό το 7% τώρα και τη λύση μπορούμε να βρούμε γι' αυτό. Σε αυτό το 7% μπορεί να είναι άστεγοι, που να μην τους ενδιαφέρει το θέμα καθόλου γιατί στην πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται έτσι κι ότι πρέπει να έχει μια διεύθυνση το άτομο, να είναι νόμιμος, να μην είναι κανένας παράνομος μετανάστης ας πούμε. Οπότε εγώ καλό θα έβρισκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να μας εξηγήσει τελικά ποιο είναι το ποσοστό της κατηγορίας αυτής την οποία θα πιάσουμε με την ε, σύσταση και ποια είναι η κατηγορία που έτσι καλώ θα μείνει απ' έξω. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο νέος πηγαίναμε στην ε, τράπεζα ή στο ταχυδρομείο, παίρναμε λεφτά, κάναμε ξέρω εγώ τι πληρωμές έπρεπε να κάναμε, αλλά δεν χρειαζόταν να ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Τώρα όμως έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκο το να χρησιμοποιεί κανείς και να διαχειρίζεται το τραπεζικό του λογαριασμό. Γιατί πρέπει να κάνει πράγματα μέσω του διαδικτύου. Είναι πιο δύσκολο δηλαδή να χρησιμοποιήσει κανείς το τραπεζικό του λογαριασμό από ότι όταν εγώ ήμουν νέος. Οπότε Μήπως θα έπρεπε να πάμε λίγο πίσω και να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την ε, προσωπική επαφή και στις τράπεζες, να μπορεί δηλαδή κάποιος να πηγαίνει στην τράπεζα και να μιλάει με τον υπάλληλο και όχι να κάθεται πίσω από τον υπολογιστή του και να τα κάνει όλα από το σπίτι. Γιατί ορισμένοι δεν τα καταφέρνουν. Όντω, υπάρχει και το άλλο, ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντα ρευστό τους κοστίζει λιγότερο. Ενώ ότι ο τραπεζικός λογαριασμός και οι διάφορες τραπεζικές συναλλαγές κοστίζουν. Όντως, Αναφέρεται παραδείγματα στην μελέτη πάντως αντικτύπου θα ήθελα κάτι πιο ξεκάθαρο για το λογαριασμό αυτών που θα παρέχει τις ε, πιο πλές, τις ελάχιστες υπηρεσίες. Γιατί όχι και να μην κοστίζει ε, κάτι τέτοιο. Σε αυτό δεν αναφέρεται όμως ή αλλιώς ε, πρέπει να λέτε ποιο θεωρείτε εσείς ότι θα είναι το ελάχιστο κόστος και να μην λέτε ένα λογικό κόστος. Ποιο θα είναι αυτό όμως. Τι θα πει αυτό ακριβώς. Και αν κάποιος δεν έχει χρήματα στο λογαριασμό του, τότε δεν γίνεται η πληρωμή. Μα ακριβώς τότε είναι που κοστίζει περισσότερο ένας λογαριασμός. Όταν δηλαδή ε, ο, αυτός που έχει το λογαριασμό δεν ε, έχει να πληρώσει και βάζει μέσα το λογαριασμό του, τότε είναι που έχει να πληρώσει τεράστια ποσά στη συνέχεια. Πάντως και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένα θέμα που θα γίνει με σύσταση. Ίσως να χρειάζεται κάποια άλλη αντιμετώπιση, νομοθεσία, κάτι άλλο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, άλλη, ο κύριος ε, Κρότσμερ, μετά Ρόσφορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντεγιόν, καταλαβαίνω τι λέτε. Και εγώ υποχρεώθηκα κάποια στιγμή να ανοίξω λογαριασμό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε καταρχάς το κόστος του λογαριασμού, Όταν δηλαδή θέλουμε να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις, θα πρέπει να είναι και εφικτές αυτές οι λύσεις, εφαρμόσιμες Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τη διακριτική μεταχείριση γιατί πολλές φορές υπάρχουν, ε, παρατηρούνται τέτοιες ε, περιπτώσεις, ε, οπότε εδώ και στους λογαριασμούς, είτε είναι πληρωμένη κάρτα είτε οτιδήποτε, να μην υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Να πηγαίνει ένας άνθρωπος στο ATM και να μπορεί να σηκώνει τα λεφτά του. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ευαίσθητο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε και γι' αυτό βασικά πήρα το λόγο. Αν θέλουμε τελικά να, κάνουμε, να επιφέρουμε πρόοδο για τους καταναλωτές, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά ακριβώς τα προβλήματα. Ο συνάδελφος Σμιτ δεν μπορεί να να παρίσταται. Μου έδωσε έτσι να διαβάσω κάτι, αλλά δεν έχει νόημα τώρα. Εγώ είπα ότι αυτά πρέπει να α, λύσουμε. Στην Γερμανία έχουμε και τα αποταμιευτικά, τις τράπεζες της ε, ε, αποταμιευτικές. Στη Γερμανία υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν τέτοιες τράπεζες. Προφανώς ε, εκεί οι υπόλοιπε τράπεζε λειτουργούν με, με το κόστος να τον αναλαμβάνει ο κάτοχος του λογαριασμού. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι που τους ε, αφορούν. Γιατί κατά τα λοιπά που τους αφορά όλο αυτό, γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα να υπάρχει ένας, ε, να ανοίγει ένας λογαριασμός ο οποίος να ε, κοστίζει πάρα πολύ. Το κόστος λοιπόν ενός λογαριασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στο φύλλο των αγγέλων. Τι εννοώ με αυτό. Ότι οι άστεγοι δεν είναι μόνη περίπτωση ανθρώπων που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Έχουν γίνει πειράματα και στη Γαλλία να θεωρούνται τα άτομα αυτά χωρίς μόνιμη κατοικία να δίνουν διεύθυνση μιας οργάνωσης με την οποία έχουν κάποια σχέση. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δύο παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, το ξέρουμε όλοι, ιδιαίτερα για τις τράπεζες. Και ξέρουμε ήδη ότι πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες αποφάσισαν να κάνουν οικονομίες και αποφάσισαν να θυσιάσουν μάλιστα κάποιους ιδιαίτερους πελάτες οι οποίοι δεν τους αποδίδουν επειδή βρίσκονται ακριβώ σε δυσκολίε. Η Μπεσεμπέ για παράδειγμα, το ανακοίνωσε και άλλε τράπεζε. Κινδυνεύουμε δηλαδή να βρεθούμε μπροστά σε μια πολιτική των τραπεζών, που είναι σε δυσκολία, που να οδηγήσει στο να βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι χωρίς να μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό, να μην τους ανοίγει τράπεζα λογαριασμό, εξαιτίας των δυσκολίων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Δεύτερον, αν πρέπει να φτάσουμε και νομίζω ότι πρέπει σε, μια, σε ένα επίπεδο ελάχιστον τραπεζικών υπηρεσιών, πρέπει να υπάρχει μια κλίδα ασφαλείας και μια κατάρτιση για το πώς να χρησιμοποιεί κανεί το λογαριασμό του. Γιατί δεν έχει νόημα να δώσουμε στους πάντες ένα λογαριασμό, αν συγχρόνω από πλευρά των τραπεζών δεν υπάρχουν κλίδε ασφαλείας. Εγώ θα ήθελα όταν ε, δεν υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό να καταργείται αντί να χρεώνεται με πρόστιμα ιδιαίτερα ψηλά για, σε, και πρέπει να τα πληρώσουν αυτά τα λεφτά άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι ισχύει όταν είναι ακάλυπτος ο λογαριασμό τους. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει και αυτή η ευαισθητοποίηση, να υπάρξει ενημέρωση και κατάρτιση του κόσμου. Τέλος, μετά την πρόταση αυτή της Επιτροπής, νομίζω και εγώ, όπως είπαν και άλλοι, ότι υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες μου κάνουν, έτσι εκ πρώτης όψεως όντως αυτός ο τραπεζικός ε, λογαριασμός πληρωμών πρέπει να έχει μια κάρτα. Να ξέρουμε ότι δεν τη δίνουν όλες οι τράπεζες την κάρτα. Επίσης, πρέπει ο λογαριασμός αυτός να συνοδεύεται και από τη δυνατότητα και διασυνοριακά να γίνονται πληρωμές. Γιατί δεν βλέπω γιατί να μην χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πρόσβαση και σε άλλη χώρα πλην της δικιάς τους. Όσον αφορά την τιμή, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να είναι δωρεάν, αν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός. Μήπως πρέπει να κρατήσουμε το reasonable price ή το minimum price, μια ελάχιστη τιμή, μια λογική τιμή. Αντίθετα, πιστεύω ότι η σύσταση δεν είναι ένα ικανοποιητικό μέσο για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Μέσα στους επόμενους μήνες είμαι περίπου σίγουρος ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο ίδιος ο Επίτροπος θα ξέρουν ότι σε 8 μήνες θα θέλουμε μία οδηγία. Άρα, εδώ είναι περισσότερο η συγκυρία που παίζει ρόλο και που θέλουμε να έχουμε κάτι εξαιτία των δυσκολιών που έχουν εκεί οι τράπεζες, αλλά αλλιώς εγώ δεν βλέπω πώς θα λυθεί αυτό το θέμα με μια σκέτη σύσταση. Αν αυτό θέλει η Επιτροπή, ε, ραντεβού σε 8 μήνες για αυτό που σας είπα. Αξίζει τον κόπο να χάσουμε το χρόνο μας για αυτή τη σύσταση στη στιγμή που έτσι κι θα κληθούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Um, thank you very much, all of you. Σας ευχαριστώ όλους. Κάποιες παρατηρήσεις να κάνω κι εγώ. Καλωσορίζω τους Φοντέιν και Νίμπλετ από την Περέκ. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να θυμηθούμε ότι κάναμε πρόταση οδηγίας, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν θέλω να καθυστερήσω και να μην βγει μια σύσταση. Νομίζω ότι μπορούμε να πιέσουμε πολιτικά και να υπάρξει γρήγορα η σύσταση. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπε η Επιτροπή, ότι στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο κάποιες τράπεζες θεωρούν ότι είναι μια καλή εμπορική ευκαιρία, ακόμα και αν στην αρχή χάνουν χρήματα, γιατί φέρνει νέους πελάτες στην τράπεζα και βλέπουν το θέμα θετικά. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα τεχνολογικά θέματα. Μιλάμε για την κινητή τηλεφωνία. Να σας θυμίσω ότι στην Ινδία σαν παράδειγμα και σε άλλες ασιατικές χώρες όπου η πρόσβαση στις τράπεζες είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχουν υποδομές καθόλου σχεδόν. Η κινητή τηλεφωνία και το ότι ο κόσμος έχει ένα κινητό τηλέφωνο με μία κάρτα SIM στην ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν cash card και είναι μια ευκαιρία για τις τράπεζες και να χρησιμοποιεί κανείς το κινητό του σαν τερματικό σταθμό και να παίρνει χρήματα. Να, τον χρησιμοποιεί σαν να έχει χρήματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί επίσης έτσι ώστε να μην είμαστε πολύ περιοριστικοί σε αυτά τα οποία προτείνουμε. Μπας περιπτώσει θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Γκέπχαρτ, ε, το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά σφιχτό. Συζητάμε με την Οικονομική Επιτροπή για τη δική του συνεισφορά και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στη συγκεκριμένη πρόταση. Είναι σαφές από τη συζήτηση που έχει γίνει ότι όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, δηλαδή και τα θέματα τα πιστοτικά και τα θέματα τα καταναλωτικά, θα πρέπει όμως η κυρία Γκέφχαρτ να κλείσει τη συζήτηση τώρα. Ευχαριστώ Μάλκομ. Σωστό είναι. Που Έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο για την πρόταση έτσι ώστε να μπορέσουμε την πρόσβαση αυτή στους βασικούς λογαριασμούς να τη διευκολύνουμε για να μπορούν όλοι οι πολίτες να κινούνται μέσα στην κοινωνία και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σωστό, είναι σημαντικό και θα παραμείνει σημαντικό ε, να, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόταση στα σημεία που δεν μπορούμε να την ε, αποδεχτούμε. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ δεν μιλούμε για την... να υποχρεώσουμε κάποιον να ανοίξει λογαριασμό. Αν δεν θέλει κάποιος ένα λογαριασμό, δεν χρειάζεται να τον ανοίξει το λογαριασμό. Αλλά την πρόσβαση στο άνοιγμα ενός λογαριασμού πρέπει να έχει. Αυτό είναι ένα δικαίωμα. Και δεν είναι το ίδιο ακριβώς, γιατί άκουσα τα σχόλιά σας ε, και ε, θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τις ε, παρανοήσεις. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να ανοίξει ένα λογαριασμό. Αν θέλει κάποιος να κυκλοφορεί μόνο με μετρητά, μπορεί να κυκλοφορεί μόνο με μετρητά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μόνο στο προσκήνιο αυτούς που τους αφορά, δηλαδή όσου όσους δεν έχουν ε, μια σταθερή κατοικία ή τους, ε, τα άτομα που δεν απολαμβάνουν ε, ε, δεν έχουν υψηλό εισόδημα. Ε, δεν μπορούμε νομίζω να βάλουμε τέτοια στεγανά. Μιλούμε και για άλλους, όπως φοιτητέ, όπως ε, ερευνητέ που ταξιδεύουν, όπως ας πούμε ε, ηλικιωμένους που θέλουν να έχουν τα χρήματα της εργασίας τους τόσα χρόνια σε κάποια άλλη χώρα, σε έναν άλλο λογαριασμό. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που μπαίνουν εδώ στο παιχνίδι και νομίζω ότι θα πρέπει να καλύπτουμε όλες αυτές τις ομάδες και να μην επικεντρωθούμε μόνο σε μία. Τα τεχνικά θέματα θα τα ξανασυζητήσουμε βεβαίως. Τι σημαίνει βασικός λογαριασμός. Σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε υπερανάληψη ή όχι. Τι είδου κάρτες μπορούν να συνδεθούν. Ε, προπληρωμένες ας πούμε πιστοτικές. τι γίνεται με άλλα ζητήματα. Ε, Αυτά μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε. Αλλά το τελευταίο που είπε, Μάλκομ, για τι δυνατότητε πληρωμών μέσω του κινητού, που είναι νέα υπηρεσία, αυτό νομίζω ότι ε, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτοί που έχουν ούτω ή άλλω πρόσβαση στο, στου λογαριασμού. Αυτό δεν είναι πρόβλημα αν θα πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού, μέσω του κινητού ή όχι. Υπάρχουν πιο βασικά θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ, πολλά προβλήματα αν αρχίζουμε να συγχαίουμε τα πράγματα. Ας περιοριστούμε λοιπόν να λύσουμε τα προβλήματα που όντως χρειάζονται λύση. Ότι δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τον λογαριασμό του, να μπορεί να κάνει ε, διασυνοριακά εμβάσματα. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι βασικός λογαριασμός και μπορεί να, είναι, ε, να τον αναλάβει οικονομικά ο πολίτης που θα τον ανοίξει. γιατί αυτό θεωρείται ουσιαστικά ε, καθολική υπηρεσία και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτό το δικαίωμα να είναι δικαίωμα που μπορεί να είναι και εφαρμόσιμο. Και εκεί, Μάλκομ, διαφωνώ μαζί σου. Δεν αρκεί η σύσταση της Κομισιόν. Και νομίζω ότι αυτό προέκυψε και από τη συζήτηση σήμερα δεν θα πάμε πολύ, ε, παρακάτω μόνο με μία σύσταση. Μια σύσταση δεν ε, καταλήγει σε τίποτα. Είναι απλά μια σύσταση. Εμείς θέλουμε κάτι που να είναι νομικό, να έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή, μια οδηγία ε, ακόμη καλύτερα, που να μπορεί να μπει στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοστεί. Μια σύσταση τι ακριβώς θα κάνει. Ούτε στην νομοθεσία θα μπει, ούτε θα αλλάξει τίποτα. Οπότε ε, δεν υπάρχει ε, λόγος, αν είναι να μιλάμε μόνο για ε, συστάσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να προσπαθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει όντως να κάνουμε κάθε προσπάθεια να προσπαθήσουμε από αυτές τις ε, προτάσει και τις συστάσεις να προκύψει μια οδηγία. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Προς το παρόν μάλλον δεν θα πω τίποτε άλλο γιατί θέλω να συνεχθώ και με τις υπόλοιπες ε, επιτροπές και θα ε, έρθω σε επαφή για την, ε, πριν την επόμενη συνεδρίαση μαζί σου για να σου αναφέρω και ποιο θα είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα αφού μιλήσω με τις υπόλοιπες επιτροπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ιβλέν. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή Νομίζω ότι η οδηγία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, ενώ μπορούμε να έχουμε εγκαίρο τη σύσταση. Αλλά, εν τώρα θα το συζητήσουμε πάλι το θέμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους και την Επιτροπή ειδικά. Ελπίζω να σας ξαναδούμε όσο προχωράει το θέμα. Περνάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για τους καταναλωτές. Για μια ακόμη φορά μετά από το φόρουμ το επιτυχές στην, στην Κρακοβία τέθηκε το, το θέμα του roaming της περιαγωγής και ο κύριος Τούν, η κυρία Τούν μάλλον έκανε μια πάρα πολύ <clears throat> ενδιαφέρουσα επίδειξη για τους νέους ε, έδειξε ότι είναι βασική προτεραιότητα για τους νέους η περιαγωγή του κινητού τηλεφώνου Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση στο παρελθόν με τον εισηγητή μας, ε, την κυρία Κόρχολα, η οποία δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα, αντικαθίσταται όμως και υποδεχόμαστε και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής για τις τηλεπικοινωνίες, ο κύριος Φοντάιν. Ξέρουμε τι είναι η Μπερέκ, αλλά να το μάθουν και αυτοί που ίσως μας ακούν και μας βλέπουν από το διαδίκτυο. Η δημιουργία της Μπέρεκ είναι προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του πακέτου Τελεκόμ. Όσοι έχετε μακρά μνήμη θα ενθυμίστε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήθελε έναν συγκεντρωτικό ρυθμιστικό ρόλο για μια τέτοια υπηρεσία. Εμείς όμως είπαμε ότι η ποιότητα και η συνεκτικότητα της ε, ρύθμισης και του διακανονισμού στα Τελεκόμ θα είναι καλύτερο με μια υπηρεσία τύπου Μπερέκ. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε σαν Επιτροπή ότι ήταν πολύ σημαντικό να μην ακούσουμε μόνο για την πρόταση για την περιαγωγή, την μελέτη επιπτώσεων α, αντικτύπου αν θέλετε της Επιτροπής, αλλά η Μπερέκ που έχει συμβουλευτικές και συντονιστικές αρμοδιότητες στα πλαίσια των νομοθετικών προτάσεων θα μας θα δώσουμε την δυνατότητα στον κύριο Φοντέιν να έρθει για πρώτη φορά σε αυτήν την Επιτροπή που ασχολείται πολύ με τα θέματα του καταναλωτή για να μας πει για τις πρόπτικες της ΜΠΕΡΕΚ στα πλαίσια του διακανονισμού της περιαγωγής. Κάτι που θα επηρεάσει τις προτάσεις που θα κάνουμε εμείς στο μέλλον. Η έκθεση έχει διανεμηθεί ήδη Έχουμε την κυρία Τούν η οποία θα δώσει ε, α, κάποιες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Ταραμπέλα εδώ. Ο κύριος Κρόιτσμαν γυμνάζεται, δεν περιάγεται προς το παρόν. Κάποιοι απόντες θα είναι παρόντες αργότερα. Εγώ θα μιλήσω για τους Βρετανούς συντηρητικούς και δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Φοντέιν για να μας κάνει τις προτάσεις του. Άκουσα με χαρά ότι εδώ μας στηρίζεται. Δεν είναι ίσως η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ. Πολύ πρόσφατα έκανα μία παρουσίαση στην Επιτροπή Ήτρε. Έχω μαζί μου τον Τζιμ Νίμπλε της Ofcom που είναι γνωστός εμπειρογνώμων στα θέματα της περιαγωγής και θα με βοηθήσει ίσως στις απαντήσεις στις πιθανές ερωτήσεις σας. Πολλές από τις παρουσιάσεις που έκανα στην Ήτρε είναι προφανώς σχετικές και με αυτήν που θα κάνω τώρα εγώ. Εδώ, όσοι ήσασταν παρόντες εκεί, τότε ελπίζω να μην βαρεθείτε γιατί υπάρχει μια κάποια επικάλυψη. Στην Επιτροπή Ήτρε παρουσίασα και τις πρώτες εμπειρίες που έχουμε με την ΠΕΡΕΚ Θα πρέπει να το δείτε αυτό αν σας ενδιαφέρει στα πλαίσια του βίντεο stream που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας. Εμείς όπως είπα θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να συλλέξουμε τις απόψεις σας στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε για την περιαγωγή είναι κεντρικό θα έλεγα ε, αντικείμενο ενασχόλησης και της ERG στο παρελθόν της προκατόχου μας και το πρόγραμμά μας το προβλέπει για το 2012. Όπως είπαμε επανειλημμένα εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά όργανα σε επίπεδο τεκμηρίωσης. Επικοινωνούμε κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή στο μέλλον. Ήδη τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύσαμε τη γνωμοδότησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον των κανονισμών περιαγωγής. Προσθέσαμε λεπτομέρειες τον μήνα Φεβρουάριο και στο τέλος του Αυγούστου εμείς δημοσιεύσαμε μια τεχνική ανάλυση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των προτάσεων της Ευρωπαϊκής. Ελπίζουμε ότι οι αναλύσεις αυτές θα συνεισφέρουν στη διευκρίνηση κάποιων θεμάτων, γιατί εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε με ε, οικονομικές λεπτομέρειες σαφέστατες τους επόμενους μήνες. Αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να σας μεταφέρω κάποια κομβικά σημεία της ανάλυσης μας, και επίσης περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς των κινητών τηλεφώνων. Οι ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι το τέλος του 2012 και ο καθένας μπορεί να έχει ένα διαφορετικό όραμα για την εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων τα επόμενα 10 χρόνια. Ξεκινώ με την ανάλυση που κάνουμε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Μπέρ εξημερίζεται γενικά την άποψη της Επιτροπής και τον στόχο της να κατεβάσει τις τιμές, να καταστήσει τις, ε, την τιμολόγηση διαφανέστερη και να επιτρέψει την ε, μια αηφόρο μορφή ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά. Αυτά τα οποία είδαμε τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια είναι ότι ο κανονισμός για την περιαγωγή ωφέλησε τον καταναλωτή, ήταν αρκετά αποτελεσματικός και έδωσε χαμηλότερες τιμές. Ταυτόχρονα έπεσαν και σχετικά γρήγορα τα διάφορα κόστη και το, το κενό ανάμεσα την τιμή όμως από τη μία και το κόστος από την άλλη είναι αρκετά μεγάλο. Πιστεύουμε ότι ο διακανονισμός που έχει προταθεί από πλευράς περιαγωγής θα είναι πάντα απαραίτητος ή θα είναι απαραίτητος για αρκετό καιρό. Όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν θα είναι αφεαυτές ιδιαίτερα ισχυρές για να καλύψουν με σωστό τρόπο τις ανάγκες των καταναλωτών και σε χονδρικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε λιανικό οι ρυθμίσεις ε, θα είναι απαραίτητες για να καλύψουν τις μεγάλες διαφορές της τιμολογήσης. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ανώτατες αυτές τιμές θα πρέπει να χαμηλώσουν στο μέλλον και να έρθουν κοντά στο κόστος, το πραγματικό και στην αντίστοιχη εσωτερική χρέωση. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί οι τιμές της περιαγωγής να φτάσουν το 2015 τις εσωτερικές τιμές όπως προβλέπεται στην ψηφιακή ατζέντα. Σε μέσες τιμές οι μειώσεις σε επίπεδο χονδρικής θα καταστήσουν ικανούς τους παροχής να προσφέρουν στους πελάτες μια ενιαία ευρωπαϊκή τιμολόγηση. Οι τιμές που θα πληρώνουν και για το roaming και για τα μηνύματα και για τα δεδομένα θα είναι πάνω κάτω αυτές που πληρώνουν και σε εθνικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά είμαστε μακράν αυτή τη κατάσταση σήμερα. Πιστεύουμε όμως ότι γενικά οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα εκεί οδεύουν. Αν μιλήσουμε τώρα για τη μεταφορά δεδομένων μέσω περιαγωγής, η πρόταση νέων ανωτάτων τιμών για το λιανικό εμπόριο είναι καλοδεχούμενες. Πρόσφατα είδαμε κάποιες πιο ελκυστικές τιμολογήσεις. Οι τιμολογήσεις αυτές όμως δεν είναι διαθέσιμες παντού. Κάποιες τιμές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν αδικαιολόγητα υψηλές. Οι ανώτατες τιμές θα καταργήσουν τις πάρα πολύ υψηλές τιμές που χρεώνονται σε πολλούς καταναλωτές στην Ευρώπη και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό ε, για την περιαγωγή σε δεδομένα. Έτσι και αλλιώ οι ποσότητες αυξάνονται συνεχώς και εναλλακτικές λύσεις όπως το Wi-Fi ε, ασκούν εναλλακτικέ πιέσει. Γι' αυτό λοιπόν οι ανώτατε τιμέ. σε αυτή τη φάση δεν θα ικανοποιήσουν απόλυτα αυτού που χρησιμοποιούν πολύ την περιαγωγή δεδομένων. Οι μέση και βαρύ χρήστε ιδιαίτερα αυτοί που χρησιμοποιούν τα smartphones, ε, ε, πράγματι έχουν ανάγκη πολύ χαμηλότερε τιμέ γιατί αλλιώς θα καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν οικονομικά να χρησιμοποιούν τα smartphone τους εφόσον πράγματι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Είναι μια παράλογη κατάσταση. Έχουν τη δυνατότητα και δεν μπορούν να την ασκήσουν. Πάντως η ζήτηση αυξάνεται όσο πέφτουν οι τιμές. Εμείς στην ΠΕΡΕΚ ελπίζουμε ότι οι εταιρείε θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του συγκεκριμένου αυτού τομέα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση από κοντά. Αν περάσουμε τώρα στις διαφορετικές λύσεις τις οποίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σαφές ότι κανένας δεν θα ήθελε να υπάρχουν μόνιμα ε, διαφθρωμένες εσωτερικές τιμές. Ούτε η Μπερέκ το θέλει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν παράλληλα με αυτές τις ανώτατες τιμές που ορίζονται θα πρέπει να αναζητηθεί μια διαφορετική λύση. Μια διαφορετική λύση που καλύπτει τις αδυναμίες της αγοράς, ενισχύει τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία απόσυρση ρυθμίσεων και διακανονισμό στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Απαιτείται μία λύση ικανή, η οποία να είναι ικανή να εφαρμοστεί γρήγορα, γιατί αλλιώς η ευκαιρία που έχουμε θα τη χάσουμε και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την αγορά θα λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους με τρόπους που δεν θα επιθυμούσαμε χαμηλότερο κόστος περιαγωγής νομίζω θα δώσει ε, κάποιες δυνατότητες στους ε, μεγάλους παροχής υπηρεσιών να βρουν σωστές λύσεις. Δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε λύσεις ακριβές στην εφαρμογή τους σε σχέση με την κλίμακα ε, πλέον εκτιμάτων τα οποία ελπίζουμε να καρποφορήσουν. Πιστεύουμε ότι μια ικανοποιητική πλήρως διαφθορτική λύση δεν έχει εντοπιστεί. Και όταν μιλάμε για ικανοποιητική, μιλάμε για μια λύση η οποία <clears throat> θα βοηθήσει και τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές ανάλογη με τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις. Εμείς μελετήσαμε πολλές διαφορετικές λύσεις στις εκθέσεις μας τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο και δεν τις βρήκαμε ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αποσύζευξη μέσω της οποίας ένας καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εσωτερικές υπηρεσίες από ένα παροχέα και τις υπηρεσίες περιογής από άλλον παροχέα χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αλλάξει το τηλεφωνάκι του. Η αποσύζευξη, το dual MC όπως λέμε, έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ότι δεν πρέπει, ότι μάλλον δεν θα εφαρμοστεί η λύση αυτή πάρα πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με την, με την ανάλυση του ανταγωνισμού, τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του να έλθουν δηλαδή οι τιμές ηλιανικές κοντά στο κόστος, είναι κάτι το οποίο γρήγορα θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό για τον καταναλωτή σύντομα. Αυτό θα επιτρέψει στους υπάρχοντες παροχείς να προσφέρουν περισσότερες ε, συζεύξεις δεδομένων πολύ πιο γρήγορα. Θα βοηθήσει επίσης και νέους παίχτες στην αγορά και στον τομέα της περιαγωγής και της λιανικής περιαγωγής όπως χρήστες ε, κινητών δικτύων ή ε, ιονί κινητών δικτύων. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα κίνδυνος και με το σύστημα Dual MC, το οποίο προτείνεται να μην είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο και να μην είναι ωφέλιμο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέτρα και λύσεις τις οποίες ε, αυτή τη στιγμή προτείνουν. Και σίγουρα το Dual MC είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και απαιτεί κόστος ε, σε σχέση με το υλικό. Εμείς ε, παρακολουθούμε τις επιλογές για την εφαρμογή της αποσύζευσης. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να ορίσουμε την καλύτερη λύση. Πάντως οι πρωτοβουλίες της βιομηχανίας να συζητήσει όλες τις επιλογές ανοιχτά και να αναζητήσει την κατάλληλη λύση είναι καλό. Επίσης θα πρέπει ο συνδυασμός λύσεων να είναι μία πιθανότητα, απλά τώρα είναι πάρα πολύ πρόημο να γίνει κάτι τέτοιο. Σαν Μπερέκ θεωρούμε ότι μία απόφαση για επιλογή ενός συγκεκριμένου μέσου εφαρμογής της αποσύζευξης θα υιοθετηθεί μόνο όταν είναι ξεκάθαρο ότι θα ωφεληθεί ο καταναλωτής και ότι τα ωφέλη αυτά θα είναι ανώτερα από το κόστος εφαρμογής και το κόστος λειτουργίας ε, του MC. Θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν αρκετά γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να στηρίξουμε ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων και να καταστήσουμε τη διαδικασία αυτή εμπορικά ενδιαφέροντα. Εμείς δεν, ε, όταν δεν έχουμε ε, θα έλεγα τη δυνατότητα να ορίσουμε σωστά ε, το εμπορικό κέρδος είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τη βιομηχανία για την ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών. Για αυτούς όλους τους λόγους, κυρίες και κύριοι, είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί ίσως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την αποσύνδεση αποσύζευξη. Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός για τις λιανικές τιμές πρέπει να παραμείνει ενισχύ, εκτός και αν αποδειχθεί, μέχρι ότου αποδειχθεί ότι οι δυνάμεις της αγοράς εργάζονται καλά. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα στις τελευταίες συζητήσεις ε, κάποιοι βουλευτές ζήτησαν οι ανώτατες τιμές να αποσυρθούν. Προφανώς συμφωνούμε μαζί τους, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ νωρίς για να το κάνουμε αυτό <clears throat> και δεν θέλουμε να διατρέξουμε οδήποτε κίνδυνο. Εάν πράγματι λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε τις ανώτατες τιμές για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να δούμε σε τι επίπεδο θα είναι αυτές οι τιμές. Και αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα να το πετύχουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει με μια στρατηγική εισαγωγή του ανταγωνισμού από την αρχή, από τη βάση. Μια τέτοια στρατηγική θα αποτύχει αν οι ανώτατες τιμές είναι τόσο χαμηλές και διώξουν ουσιαστικά τους βασικούς εμπλεκομένους ε, στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Από την άλλη, οι ανώτατες τιμές δεν θα πρέπει να είναι τόσο υψηλές, οπότε να μην προστατεύουν σε καμία περίπτωση τον καταναλωτή. Εδώ λοιπόν είναι δύσκολο να βρούμε μια καλή ισορροπία και δεν υπάρχει καμία επιστημονική μέθοδος να μας βοηθήσει. Κατανοώ λοιπόν τις δυσκολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, σαν Μπέρεκ, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία ισορροπία, να χαμηλώσουμε τις προτάσεις από το 2014 για ανώτατες τιμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι ένα λιανικό περιθώριο κέρδους 200% σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τρεις φορές πάνω από το κόστος. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την είσοδο στην αγορά νέων παικτών και ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όσο αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός οι καταναλωτές είναι προφανές ότι λόγω των χαμηλών τιμών θα προστατεύονται καλύτερα. Λόγω όλων αυτών των αβεβαιοτήτων και λόγω του μακροπροθέσμου προγράμματος το οποίο έχουμε μπροστά μας πρέπει να πούμε ότι μια αναθεώρηση το 2015 όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει τη δυνατότητα να επανεξετάσουμε τη στρατηγική μας θα πρέπει να προβλέπεται στον κανονισμό η επαναξιολόγηση. Πρώτον θα πρέπει να ελέγξουμε σε ποιο βαθμό οι δυνάμεις της αγοράς μέχρι τότε κινητοποιήθηκαν από τα διαφορετικά μέτρα ή όχι και πόσο έχουν επηρεάσει τις τιμολογήσεις για όλες τις μορφές παροχής υπηρεσίας. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό οι προσδοκίες σχετικά με το κόστος έχουν εκπληρωθεί. Δέκα χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για την ισχύ μέσων παρέμβασης στις λιανικές τιμές. Και σαν ρυθμιστικές αρχές εμείς εξετάζουμε τις αγορές μας κάθε δύο με τρία χρόνια και το πλαίσιο, νομίζω το χρονικό εδώ είναι αρκετά καλό. Και τρίτον, η ανάγκη συνέχισης της επιβολής των συγκεκριμένων αυτών λιανικών τιμών, ανωτάτων τιμών, η σχέση των τιμών αυτών με το κόστος των χονδρικών τιμών και το κόστος της παροχής υπηρεσίας είναι θέματα που πρέπει να επανεξεταστούν. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω τώρα για κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται σαφώς στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε για τη συμπερίληψη και σας απασχολεί και εσάς αυτό, του εξής. Θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν το 2010 σχετικά με την περιαγωγή δεδομένων θα πρέπει να διευρυνθούν και για τη χρήση τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο τεχνικά να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει αρκετή προσπάθεια. Τα μέτρα τα οποία εισήχθησαν πράγματι αφαίρεσαν και απομάκρυναν κάποιες φρικτές ιστορίες καταναλωτών που πλήρωναν χιλιάδες ευρώ χωρίς να χρησιμοποιούν πάρα πολύ τις υπηρεσίες. Παρ' αυτά είναι υψηλές οι τιμές αναμονάδα και δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης μείωσης. Κάποιες εταιρείες όμως ήδη έχουν εφαρμόσει κάποια τέτοια μέτρα σε εθελοντική βάση περιορισμού του κόστους Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τη μείωση τους κόστους για τους καταναλωτές εντός αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα μέτρο εσωτερικής αγοράς γιατί παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές από υπηρεσίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη προς πολίτες οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρώπης. Και γι' αυτό κλείνοντας κυρίες και κύριοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ΠΕΡΕΚ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των μεγάλων χρηστών και των μεσαίων χρηστών και των ε, μικρών σε εισαγωγικά χρηστών. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε σαν στόχο να βρούμε μια διαφθορτική λύση η οποία είναι ο βασικός μας στόχος μια διαφορετική λύση που θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο στην αγορά περιαγωγής μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιομηχανία και όλους τους άλλους εμπλεκομένους. Μέχρι ότου γίνει αυτό όμως και αν δεν υπάρξει μια διαφορετική λύση η οποία αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει το θέμα της μείωσης των τιμών με αποτελεσματικό τρόπο, τότε θα πρέπει να παραμείνουν οι ανώτατες λιανικές τιμές. Θεωρώ, ιδιαίτερα όταν μιλάω σε εσά, ότι εμείς σαν Μπερέκ είναι ξεκάθαρο ότι θα σας δώσουμε κάθε τεχνική, τεχνολογική λεπτομέρεια και τεκμηρίωση που θα έχετε ανάγκη στις συζητήσεις σας. Well, thank you very much indeed, uh, for... Ευχαριστώ. Βλέπετε νομίζω γιατί ήταν τόσο σημαντικό να έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Μπερέκ. Εσείς είσαστε ο πρόεδρος του Ολλανδού ρυθμιστή, ταυτόχρονα είσαστε και πρόεδρος της Μπερέκ. Λοιπόν, έχουμε μισή ωρίτσα για ερωτήσεις. Ο κύριος Τέλεβαχ είναι εδώ, που παρουσίασε και την αξιολόγηση επιπτώσεων της ε, Κομισιόν, είναι παρόν, οπότε αν θέλει μπορεί να επανέλθει. Βεβαίως τα έχετε ξανακούσει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αν έχετε οτιδήποτε να μας ε, πείτε, χρήσιμο θα είναι. Και επίσης, στην τελική, τελευταία σας πρόταση για, το, για το, την περιαγωγή εκτός α, Ευρώπης. Η Επιτροπή ε, υπέβαλε την πρόταση για, την, για το περιορισμό των ορίων περιαγωγής, του κόστου περιαγωγής εκτός Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς. Οπότε γνωρίζουμε το θέμα αυτό, σε αφορά και την ενημέρωση των πολιτών ε, με τα SMS που λαμβάνουν όταν μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Είναι λοιπόν αρκετά καινοτόμο η προσέγγιση. Βεβαίω κάποια τεχνικά, διαρθρωτικά θέματα αφορούν περισσότερο την Επιτροπή βιομηχανία, Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και αυτά. Λοιπόν, η κυρία Τιούν έχει το λόγο και μετά η κυρία Κόρχαλεκ εκ μέρου της, του Mrs. Corolla regrets uh, she cannot be here. Η κυρία Κόρχολα λυπάται που δεν είναι παρούσα, αλλά δυστυχώ έχει μια άλλη ανηλυμένη υποχρέωση. Έπρεπε να είναι στη Φιλανδία. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά σημεία που μου έχει δώσει θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Αυτό που λέει λοιπόν η κυρία Κόρχολα είναι ότι η περιεγωγή είναι ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα το οποίο άπτεται πολλών, ε, πλήττει μάλλον πολλούς ε, καταναλωτές και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι αναλύσει δείχνουν ότι ο προηγούμενο κανονισμό, για το κανονισμό, ο πρώτο και δεύτερο, για, το, για την παραγωγή έφερε πολλά ωφέλη. Αλλά η αγορά δεν έχει αλλάξει πολύ έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει μια, μια μόνιμη λύση για την περιαγωγή. Τώρα που κυκλοφορούν και τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones και έχουν πολλές ε, εφαρμογές αλλά υπάρχουν πολύ, και πολύ περισσότερα βιομηχανικά μοντέλα και όλα αυτά γίνονται με πολύ ταχύς ρυθμούς, πρέπει και εμείς να είμαστε ταχύς ώστε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ανταγωνισμό θα μειώσει τι ε, τιμέ περιεγωγή. Η κυρία Κόρχολα θεωρεί ότι θα γίνουν πολύ ωραίε συζητήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να θυμίσει τη σημασία να ολοκληρωθεί όλο αυτό, όλη αυτή η δουλειά σχετικά άμεσα, ώστε να μπορέσουμε σε πρώτη ανάγνωση να έχουμε τελικά συμφωνία. Να ρωτήσω εγώ εδώ δύο πράγματα. Είναι πολύ βεβαίω οι προτάσεις, αλλά θα ήθελα να πω ότι οι τιμές ελληνικής για την ε, πυραγωγή δεδομένων είναι πάρα πολύ υψηλές. Τώρα το περίπου το, το όριο είναι 300, για τη Λενική είναι 300% της χοντρικής. Προφανώς είναι πάρα πολύ αυτό, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Στις εθνικές αγορές είναι περίπου 30 με 40%. Και υπάρχει στα πλαίσια αυτά έτσι ένα περιθώριο ανταγωνισμού. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να άρουμε αυτούς, τους, αυτά τα ανώφλια. Νομίζω ότι πρέπει να το μελετήσουμε πιο πολύ και να δώσουμε χρόνο στην αγορά για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Και αυτό που χρειάζεται είναι να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να ξέρουν ότι οποτεδήποτε δουλεύουν σε εξωτερικό ή σπουδάζουν δεν θα πληρώνουν πολύ ψηλότερες τιμές από αυτές που θα πλήρωνε να έμεναν στη χώρα τους. Το βασικό σημείο είναι ότι η κλίση, η κρίση του ίντερνετ ή η, τα, τα, η αποστολή μηνυμάτων θα πρέπει να είναι ε, πάρα πολύ ευθυνή, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ ακριβή, μόνο και μόνο επειδή άλλαξαν χώρα. Μια που ούτως ή άλλως τώρα σύνορα πλέον δεν υπάρχουν. Η αποσύνδεση λοιπόν και για το GLMC που είπατε, ε, αυτή η λύση δεν είναι νομίζω επαρκή. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα αυτό. Αλλά ίσως θα έπρεπε να δούμε και άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, ε, για παράδειγμα περιεγωγή όπως στην χώρα του καθενός. Ας πούμε εθνική ταρίφα συν ε, ε, ποσά ανάλογα με το κόστος, ανάλογα με την κατανάλωση. Ε, νομίζω ότι αυτή η επιλογή είναι η πιο κοντινή σε αυτή ε, το, στόχο της ψηφιακή ατζέντα. Ίσως η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο και οι αρμόδιοι θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια μελέτη, γιατί δεν έχουμε κάνει μια μελέτη που να μας δείχνει πώς θα επηρεάσει αυτό την αγορά, γιατί στην αξιολόγηση επιπτώσεων περιγράφει λίγο ακροθυγός όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι έτσι υπήρξαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία. Ίσως να ήταν μισή σελίδα, μισή σελίδα για το, για το θέμα αυτό. Ενώ ε, η αποδέσμευση αναφέρεται λεπτομερέστατα σε πολλά σημεία. Οπότε, ε, ερώτημα. Η Μπέρεκ τι άποψη έχει για αυτό το Rome Like at Home. Ευχαριστώ. Um, Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει να παρέμβει κάποιο για του ε, ε Ο κύριο Κρότσμαν είναι σίγουρα εδώ, οπότε μπορεί να μα μιλήσει. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφο. Δεν, ε, είναι σαν να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε τις τεχνικές ε, προϋποθέσεις. Έτσι συμπεριφερόμαστε να πάει κανείς δηλαδή να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του στο εξωτερικό χωρίς να πληρώνει πανύψηλα, πολύ ψηλό κόστος ε, περιαγωγής. Το κόστος, ε, ναι, προφανώς ε, υπάρχει, αλλά θα πρέπει να υπολογιστεί σωστά. Το ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα να θέσω εγώ. Ε, ήσασταν και εσείς αρκετά επικριτικό στην παρέμβασή σας. Ε, είπατε ότι τελικά δεν είναι όλα πολύ εύκολα σε τεχνικό επίπεδο. Ερώτημα, αν τελικά κάτι δεν λειτουργεί ε, σε μια πιο ε, σύντομη περίοδο και αν δηλαδή χρειάζεται δύο-τρία χρόνια για να λειτουργήσει, αυτά τα δύο-τρία χρόνια ποια εναλλακτική έχουμε. Υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικέ λύσεις. Μήπως πρέπει να συζητήσουμε αυτές τις εναλλακτικέ έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτά τα κόστη να τα μειώσουμε. Γιατί εδώ μιλούμε και για ε, ίντερνετ, ε, χρήση του ίντερνετ από το τηλέφωνο, δεν μιλούμε μόνο για μια απλή κλίση, μιλούμε δηλαδή για μεγάλες, ε, μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Οπότε ε, αυτέ θα πρέπει να φροντίζουμε να μην συνοδεύονται και από υψηλά κόστη. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σάγκστρομ. Ευχαριστώ. Ε, βασικά συμφωνώ με τους τρεις προλαλήσαντες γιατί και εγώ νιώθω ότι ναι, χρειαζόμαστε ρύθμιση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εσωτερική αγορά. Ε, συμφωνώ επίσης, παρόλο που δεν ξέρω λίγο για τη διάρθρωση, αλλά αναρωτιέμαι πόσο θα κοστίζει η εφαρμογή όλων αυτών. Ε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να χρειαστεί χρόνο να το ξέρουμε. Έχω λοιπόν τι αφιβολίε μου, τι επιφυλάξει μου. Πάντω, το πιο σημαντικό για μένα είναι οι διαφορέ στι τιμέ. Και ιδιαίτερα οι τιμέ χονδρική είναι πολύ σημαντικό. Και στη Λιανική βέβαια να μην φορτώνεται υπερβολικό κόστος ο καταναλωτής. Το έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή μας πάντως. Ως Σουηδός έχω φίλους που δουλεύουν για μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Η παραγωγή για ένα γιγαμπάιτ, το πρώτο μου, έτσι, Καλά, μην μιλάμε για megabytes, γιατί μετά υπάρχουν πάρα πολλά μηδενικά και μπερδευόμαστε. Το gigabyte είναι πιο ρεαλιστικό. Μισό gigabyte συνήθως είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι η παραγωγή στοιχίζει κάτω από ένα ευρώ, κάτω από ένα δολάριο για ένα gigabyte. Οπότε 10 ευρώ το gigabyte είναι πάρα πολύ λογικό. Και έτσι οι υπάροχοι έχουν μεγάλο περιθώριο και μπορούν να επενδύσουν και για παραπάνω δυνατότητες. Αυτό δηλαδή που έχει σημασία στη ρύθμιση είναι να φτιάξουμε μια πραγματικά εσωτερική αγορά όπου οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους χωρίς να το σκέφτονται ότι έχουν αλλάξει χώρα, χωρίς να τους νοιάζει. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε να επενδύσουν ε, οι πάροχοι σε νέες υποδομές εφόσον χρειάζεται. Πάντως εφόσον κοστίζει η παραγωγή κάτω από 1 ευρώ, 10 ευρώ είναι υπεραρκετό. Μου φαίνεται πολύ λογικό. Τότε είχαμε πει 20 ευρώ για τη Λιανική. Είναι συζητήσιμο πάντα. Τι θα λέγατε εσείς για αυτά τα επίπεδα περιαγωγής, αυτά τα επίπεδα τιμής. Πρόεδρος. Και η κυρία Κέπαρτ θέλει το λόγο, αλλά και εγώ θέλω να μιλήσω εκ μέρους της ομάδας μου. Από αυτό που είπατε στο τέλος, μια λύση για να βοηθούμε τους καταναλωτές να μπορούν με περιαγωγή να μιλάνε εκτός Ευρώπης χωρίς να τους νοιάζει. Ίσως αυτό πρέπει να προτείνουμε ως Επιτροπή. Αυτό το θέλει ο πολίτης. Έρχομαι τώρα στο γενικότερο θέμα. Συμφωνώ με την προσέγγιση τη δικιά σας. Τα διαρθρωτικά μέτρα δεν έχουν αναλυθεί και αναπτυχθεί επαρκώς όσο θα έπρεπε τουλάχιστον. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνει. Δεν είναι δικιά μας βέβαια δουλειά ε, η τεχνολογία, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για τον έλεγχο των τιμών και να μπορέσουμε να κρίνουμε σωστά ανάλογα στη συνέχεια να γίνουν και επενδύσεις. Εσείς είσαστε πιο κοντά στην αγορά, οπότε δικές σας προτάσεις μπορεί να δίνουν στους παρόχους λιγότερα περιθώρια, οπότε εμείς ευχαρίστως να σας ακολουθήσουμε. Αυτή νομίζω ότι θα είναι γενικά η του Κοινοβουλίου. Για το θέμα των δεδομένων, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι Υπάρχουν διάφορα σχέδια για δεδομένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μάλιστα για την χρήση των δεδομένων που φαίνονται πολύ ελκυστικά στον κόσμο. Οι συνάδελφοι αγοράζουν τέτοιες υπηρεσίες. Μια υπηρεσία πανευρωπαϊκών δεδομένων λοιπόν υπάρχει. Ίσως για αυτούς που έχουν και iPad ή που έχουν δύο κινητά. Πάντως τέτοια εργαλεία που χρησιμοποιεί κανείς όταν ταξιδεύει, σίγουρα θα μας κατακλείσουν όλο και περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν και ένα πρόγραμμα σταθερού κόστους. Προς τα εκεί πάει η αγορά των καταναλωτών. Πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι η ρύθμιση δεν εμποδίζει τους παρόχους να προσφέρουν πακέτα τιμών στους καταναλωτές. Δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό. Να ενθαρρύνουμε εμείς τον ανταγωνισμό. Αλλά σίγουρα πριν καταλήξουμε σε μία μόνιμη λύση θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος δοκιμής. για το Dual MC. Άκουσα τις επιφυλάξεις σας. Βλέπουμε ότι οι πάροχοι καλύπτουν ε, τα δίκτυα με τιμές χοντρικής πολλές φορές. Αναφέρετε κι εσείς στην παρουσίασή σας πώς έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι, για παράδειγμα, άμα μπουν σε ένα ξενοδοχείο που δεν έχει Wi-Fi, τι κάνουν, πληρώνουν σε μια εταιρεία για να έχουν πρόσβαση. Λύσεις δηλαδή υπάρχουν πολλές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς πολύ προσεκτικοί όταν προσπαθούμε να δώσουμε συνταγές. Με αυτό το πακέτο περιαγωγής, πάντως, νομίζω ότι καλύπτουμε τα συμφέροντα όλων. Και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε μια διαρθρωτική λύση. Ξέρουν ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, αλλά δεν υπάρχει επιχείρημα για την αναγκαιότητα, οπότε αυτό που προσφέρουμε εμείς στους καταναλωτές είναι πολύ σημαντικό πρέπει να δούμε συγχρόνως πώς θα λειτουργήσουν οι άλλες πτυχές του πακέτου όταν πηγαίνουν οι πολίτες σε άλλη χώρα και ε, εκεί ε, τους στέλνουν κάποια δεδομένα ώστε το πακέτο μας τελικά να είναι πραγματικά προσανατολισμένο στον καταναλωτή και ο καταναλωτής να μπορεί να αποφελείται από τις νέες τεχνολογίες. Αυτά είχα να πω εγώ. Τώρα, Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Η κυρία Κέπαρτ, ο κύριος Δεκάμπος, ο κύριος Δεγιόγκ. Είστε σκιώδης. Α, γιατί αν είσαστε, συγγνώμη που σας άφησα απ' έξω πριν. Θα επιτρέψετε στην κυρία Γκέπαρτ πρώτα και μετά εσείς. Ε, Ευχαριστώ. Ήδη υπόθηκαν πολλά, οπότε δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Δύο πραγματάκια μόνο θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτές οι ε, ιονοί υποδομές που είπατε, αυτά τα virtual structures, θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς είναι, γιατί πάντα έχω έτσι μια δυσκολία όταν αφήνουμε την πραγματική οικονομία. Είδαμε τι σημαίνει αυτό για τις ε, χρηματαγορές. Ε, θέλω να καταλάβω εδώ τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα virtual structures και επίσης θα μπορούσατε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε με, αυτή την, ε, με το λιανεμπόριο, μας είπατε το τυχονδρική που μπορεί να απολυθεί διασυνοριακά οι υπηρεσίες. Ε, δεν το κατάλαβα. Αλλά Θέλουμε προφανώς να ανοίξουμε νέες αγορές, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε και τους καταναλωτές, οπότε θα ήθελα έτσι λίγο περισσότερα πράγματα να μου πείτε. Το δεύτερο, κάτι που δεν υπόθηκε από κανέναν μέχρι στιγμής, ή τέλος πάντων το άκουσα, στα χρόνια που έχουμε κάνει όλη αυτή τη συζήτηση, μιλήσαμε για την ευθύνη και την υπευθυνότητα των εταιριών, κυρίως αυτών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά συμπεριφέρονται σαν να είναι εθνικές οντότητες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ είναι ο συνάδελφος Κοράγια Δεκάμπος. Ας πούμε ότι έχει ένα συμβόλαιο σε μία ε, σε ένα πάροχο στην ε, Πορτογαλία, εγώ στον ίδιο πάροχο στην ε, Γερμανία και εδώ στο Βέλγιο μιλούμε και οι δύο στο τηλέφωνό μας. Παρόλο που έχουμε τον ίδιο πάροχο και έχουμε υπογράψει την σύμβαση με τον ίδιο πάροχο και οι δύο πρέπει να πληρώσουμε περιεγωγή και μάλιστα υψηλά, υψηλό τέλο για την περιαγωγή. Πώ δικαιολογείται αυτό, αυτό το θέμα πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γιατί πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αν α πούμε ο ένα με τον άλλον ε, έχει διαφορετικό πάροχο, εντάξει, ίσω να μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά αν είμαστε στην ίδια εταιρεία, στον ίδιο πάροχο, πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η κερδοσκοπία. Γιατί εκεί ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι εταιρείε είναι ότι εκμεταλλεύονται τις εθνικές τους υποδομές. Οπότε θα ήθελα αυτές οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται ευρωπαϊκά να, να αναλάβουν και την ευθύνη που τους αναλογεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η απόψη σας προς αυτό. That's true. Of course, you do have an uh, in your own countries, which... Μα έχετε και λογαριασμό στη χώρα σας που τον πληρώνετε με το ίδιο νόμισμα. Ίσως να είναι το πακέτο που έχει ο κύριος Κάμπο, ε, ε, Κάμπος, διαφορετικό από το πακέτο που έχετε εσείς. Ο κύριος Δεγιόγκα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σκιώδης εισηγητής ή δεν είμαι. Να σας πω την αλήθεια. Ε, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, βλέπετε, στην ΚΟΕ, μια που η κυρία Σβένσον δυστυχώς αποχώρησε. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα ξαναδούμε όλους τους καταλόγους και θα ξέρουμε ποιος εκπροσωπεί τι και ποιος κάνει τι και ποιος είναι σκιώδης. Πάντως ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά περίεργο όταν έρχομαι από την Ολλανδία και έρχομαι εδώ στις Βρυξέλλες, περνάω κάποια σύνορα και μιλάω πιο ακριβά στο τηλέφωνο από ότι αν πάω από ένα σημείο της Ολλανδίας σε ένα άλλο σημείο της Ολλανδίας. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη, δηλαδή περισσότερα χιλιόμετρα. Αν δηλαδή οι τιμές αλλάζαν ανάλογα με την απόσταση θα το καταλάβαινα. Ενώ το να μιλάει κανείς πιο ακριβά επειδή αλλάζει χώρα δεν το καταλαβαίνω. Επειδή περνάς κάποια σύνορα πρέπει να πληρώνεις πιο ακριβά αν και είσαι πιο κοντά είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω και δεν το βρίσκω αρκετά ευρωπαϊκό. Εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έπρεπε να υπάρχει μία ταρίφα και όχι πολλές. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Φοντέν. Βλέπετε, η Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και όντως ο κόσμος είναι ευγνώμων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που έκανε για την περιαγωγή. Πάντως το βασικό είναι να τα βλέπουμε τα αποτελέσματα στην αγορά. Τι πιστεύει ο κύριος Φοντέν ότι είναι εφικτό όσον αφορά τον ανταγωνισμό και πότε μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Έπειτα υπάρχουν και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Αν υπάρχει ένα τομέα που είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και δύσκολος για να πάρει αποφάσεις ο καταναλωτής, είναι ακριβώς οι τηλεπικοινωνίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνει και να διαλέξει ανάμεσα στις προσφορές που του γίνονται. Μήπως λοιπόν και εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερη διαφάνεια. με μια πρόταση που να αποσυνδέει για παράδειγμα την ε, περιαγωγή από τα εθνικά πακέτα ή θα γίνει ακόμα πιο περίεργο το πράγμα και πιο περίπλοκο. Πάντως, καλό θα ήταν να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για τον καταναλωτή και να μπορεί αυτός να επιλέγει πιο εύκολα το πακέτο που θα πάρει. Κάτι άλλο, πάλι που με αφορά ως καταναλωτή άμα θέλω να πάρω μια νέα συνδρομή, διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή για τη μεταβίβαση δεδομένων. Μου είπαν, αν είσαστε επιχειρηματίας, ίσως θα μπορούσαμε να σας δώσουμε ένα επιχειρηματικό πακέτο, πολύ πιο φτηνό. Ε, είμαι επιχειρηματίας όμως, αφού έχω να βοηθώ εδώ. Δεν είμαι. Χρησιμοποίησα λοιπόν αυτό το καθεστώς και κατάφερα και πήρα ένα πιο φθηνό πακέτο επιχειρηματία. Μα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όμως τα πράγματα, λοιπόν τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Thank you very much. Well, I remind you that we did a lot of work on contract Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά στο θέμα του πακέτου για τις καθολικές ε, υπηρεσίες, όπως επίσης και για τις ρυθμίσεις των συμβάσεων. Παρακαλώ από τους συναδέλφους να είναι πάρα πολύ σύντομοι. Υπάρχουν τρεις συνάδελφοι που περιμένουν το λόγο. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. ο κύριος Κορέιρα Ντεκάμπος σε μία μη κορεσμένη αγορά η αγορά μπορεί να δεχθεί εισερχόμενος. Υπάρχουν πλέον εκτήματα οι νεοεισερχόμενοι ανεβαίνουν στο επόμενο επίπεδο γρήγορα, ωφελούμενοι οικονομικά και από το ανώτατο αυτό όριο τιμών. Η κατάσταση αυτή είναι λίγο άδικη βέβαια. Η απόφαση για το roaming που ελήφθη το 2004 ήταν μια απόφαση που επηρέασε όλους τους Ευρωπαίους και περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα. Είπατε ότι τεχνικές διαφορετικές λύσεις σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο να βρεθούν. Εάν όμως η αγορά είναι σε θέση να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο, γιατί να μην έχουμε επίσης μια χρονική διάρκεια συγκεκριμένη για τις ανώτατες τιμές με ε, συγκεκριμένες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τις ανώτατες αυτές καθορισμένες τιμές, αλλά μειούμενες σαν τάση λόγω του περιθωρίου, με συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου, ορισμένου χρόνου κάθε ε, καταναλωτής θα γνωρίζει εκ των προτέρων ότι μπορεί να αλλάξει τον παροχέα του πάρα πολύ γρήγορα και η εταιρεία θα γνωρίζει επίσης ότι το συμβόλαιο και αυτό πρέπει να αλλάζει. Ξέρω ότι αυτό δημιουργεί πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά θα ωφελήσει ιδιαίτερα τον καταναλωτή. Δεν γνωρίζω όλες τις τεχνικές δυσκολίες για μια τέτοια προσπάθεια, αλλά θα ήθελα την τη γνώμη σας γι' αυτό. η κυρία Σάλντε Μόζε, μετά η κυρία Μπίλτ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν εργαζόμαστε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σαν στόχος μας είναι να μην υπάρχουν διαφορές σημαντικές στην εσωτερική αγορά. Μιλάμε για ενιαία αγορά και αυτό πρέπει να φαίνεται και στην τιμολόγηση του roaming. Θα πρέπει λοιπόν να το υπογραμμίσουμε αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Μιλάμε για ανώτατες ορισμένες τιμές, για, το, για την κερδοφορία των επιχειρήσεων κτλ. Αλλά εμείς βλέπουμε το αντίθετο εδώ. Βλέπουμε ότι επιτρέπουμε εμείς με τα μέτρα μας να υπάρχουν τέτοιου είδους πολύ σημαντικές διαφορές στις τιμές. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες διαφορές ανάλογα με το που ζει ο καθένας. Ε, μία ερώτηση λοιπόν. Δεν έχει τεθεί το θέμα αυτό πάρα πολύ ακόμα. Εξακολουθούμε να βλέπουμε όμως παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε μεθοριακές περιοχές, στα σύνορα ας πούμε Γερμανίας-Δανίας, και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τους λογαριασμούς τους γιατί δεν συνειδητοποιούν ότι στην ουσία βρίσκονται σε περιαγωγή όταν ομιλούν με το τηλέφωνό τους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα πρέπει οι πολίτες παράνομα και άδικα να υφίστανται τέτοιου είδους χρεώσεις. Πείτε μας αν έχετε λύσεις για τέτοιου είδους καταστάσεις. Ευχαριστώ η κυρία Μπίλτ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο κόσμος σε σχέση με την ψηφιακή αγορά είναι το κόστος του roaming. Ανησυχούσα λίγο για τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τις ανώτατες αυτές τιμές, τις λιανικές. Αυτό προστατεύει τους καταναλωτές, αλλά η διαφάνεια και η ελευθερία είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των καταναλωτών. Η ελευθερία και η επιλογή θα βοηθήσει τον καταναλωτή. Ας μην είμαστε τόσο περιοριστικοί, ας αφήσουμε ελεύθερη την αγορά. Και το να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το 14 διαφορετικά μέτρα, και το λέω προς την Επιτροπή αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Ελευθερία θέλει ο καταναλωτής και αυτό θα μειώσει και το κόστος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε την ισορροπία αν θέλετε, αφαιρώντας τις ανώτατες τιμές επιτρεπόμενες από τη μία και καινοτομώντα από την άλλη. Και τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί όσο έχουμε πάντα ανώτατες τιμές εμποδίζουμε τις εταιρείες να χαμηλώσουν τις τιμές τους και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάτσι 22. Um, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Δεν βρίσκομαι απλώς ανάμεσα στους δύο συναδέλφους, αλλά και η παρότησή μου είναι ανάμεσα στους δύο συναδέλφους πολιτικά. Γι' αυτό το wholesale cap που είπατε βρίσκεται πάνω από την τιμή που τελικά πληρώνεται από τους ε, χονδρεμπόρους. Αυτό δεν δείχνει ότι υπάρχει χώρος για περισσότερο ανταγωνισμό. Ε, Η κυρία Ναι, ε, για τις περιφερειακές ε, περιοχές θα ήθελα εγώ να μιλήσω. Ας πούμε στην Ελβετία είχα μια τέτοια εμπειρία. Η πάροχοι ε, ουσιαστικά αυτός που έχει το, το πιο ισχυρό σήμα προσπαθεί να ε, υπερκαλύψει όλους τους υπόλοιπους και να ε, προσελκύσει τους ε, πολίτες που ζουν σε αυτές τις συνοριακές περιοχές. Νομίζω ότι αυτό είναι αφέμητο ανταγωνισμός. Και επίσης αυτό που είπε η συνάδελφος για τον όγκο εγώ είμαι σε έναν πάροχο που λέει ότι τώρα στο εξωτερικό προσφέρει ό,τι απεριόριστο ίντερνετ ας πούμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι για μια εβδομάδα εγώ έχω 50 MB ε, δικαίωμα να, να χρησιμοποιήσω, αλλά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ε, email, ας πούμε, να στείλετε ή να διαβάσετε, ε, σε δύο-τρεις μέρες τελείωσε. Τα, έχεις χρησιμοποιήσει τα 50 MB, και νομίζω ότι το θέμα αυτό σχετικά με τον όγκο και τις τιμές που επιβάλλονται είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευχαριστώ. Ίσως όντως αυτό να είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Η κυρία Μπίλντ έχει κάνει πολλή δουλειά για την λιανοπόληση, ε, για το λιανικό εμπόριο. Ας ακούσουμε τώρα τον κύριο Φοντέιν να μας απαντήσει σε όσο χρόνο μας έχει απομείνει. Όλα, πρόεδρε, θα... Έχουμε και την και αντίτυπα της ε, εκθεσής σας, οπότε ε, Βεβαίω, αν θέλετε να απαντήσετε, ευχαρίστω να σα ακούσουμε. Βεβαίω, βεβαίω, πρόεδρε, ευχαρίστω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα ερωτήματα. Αν δυσκολευτώ, θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφο. Κυρία του, ο ανταγωνισμό, ναι, θα μειώσει τι τιμέ. Όντω, αυτό είναι, αυτή είναι και η δική μα επιθυμία οι τιμέ τη Λιανική είναι πολύ υψηλέ. συμφωνούμε επίση, και αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα τη έκθεση από τα πορίσματά τη. Αυτό που προτείνεται είναι το γιατί τα, δεν μπορεί να μεταφέρονται τα περιθώρια που υπάρχουν και, στο και στη διασυνοριακή περιαγωγή. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαφορά στο κόστο ω προ αυτό, αλλά θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε όσο όλο το περισσότερο ανταγωνισμό στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να υπάρξουν η ισορροπία ε, μεταξύ του κόστου στο εξωτερικό και του κόστου στην εθνική αγορά. Ε, θα πρέπει όντω να φτάσουμε τον ε, στόχο, θα πρέπει όμω να μειώσουμε και την τιμή σύντομα. Κύριε Κρόιτσμαν, η κριτική για τις διαρθρωτικές λύσεις, συμφωνώ. Και εμείς είμαστε πολύ σκεπτικοί, αλλά πιστεύω ότι συμφωνούμε σε πολλά πράγματα και ένα από αυτά προκύπτει σε, πολλά, σε πολλές παρεμβάσεις σας ότι δεν θα πρέπει να έχουμε για πάντα ρύθμιση τιμών. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Καμία βιομηχανία ε, για τα επόμενα 10-20 χρόνια, ας πούμε, δεν θα πρέπει να προστατεύει, να την χάνει προστασία σε επίπεδο τιμών. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια φυσιολογική αγορά, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτόν τον δρόμο και τελικά να καταλήξουμε σε μια φυσιολογική αγορά. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα πρέπει απλώς να έχουμε την ίδια τιμή παντού. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα, έχει, θα υπάρχει ρύθμιση τιμών για πάντα. Ε, εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά οποιαδήποτε πολιτική άποψη και να έχει κάποιος, αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα βοηθούσε. Κυρία Έγκστρομ, για τις διορθωτικές λύσεις που προτείνονται έχετε κάποιες αμφιβολίες. Ερωτήσατε κάτι για τα δεδομένα και για, τις, ε, για τα επίπεδα τιμών που έχουμε ε, προτείνει. Θα ήθελα ο συνάδελφος να το σχολιάσει αυτό. Γενικώ, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν για τις ανώτατες τιμές βασίστηκε στην ανάλυση που έχει κάνει η Μπέρεκ κατά πολύ. Οπότε δεν νομίζω ότι εμεί θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό που προτείνονται. Αλλά για το, τουλάχιστον για το χοντρεμπόριο. Αλλά δύο πράγματα θέλω να πω. Οι NRS εντωμεταξύ δεν έχουν ξανακάνει ε, ανάλυση για τις τιμές που... και δεν έχουν ε, ρύθμιση για τις εθνικές αγορές, οπότε δεν έχει υπάρξει ανάγκη να μπούμε σε αυτό το θέμα του κόστους. Ε, το κάνουμε βέβαια, αυτή τη δουλειά τώρα την κάνουμε, αλλά οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή είναι έτσι πολύ πρόωροι, πολύ προκαταρτικοί. Οπότε όταν θα έχουμε καλύτερα μοντέλα κόστους για όλη την Ευρώπη θα είναι πιο κοντά οι υπολογισμοί μας σε αυτά που πρότεινε ο κύριος Έγκστρομ. Ε, ε, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώ ό,τι αφορά την ανάλυση των, ε, του μοντέλου κόστου που προ το παρόν κάνουμε. Τώρα, το θέμα με τι ανώτατε τιμέ είναι η σχέση μεταξύ ε, τη ανώτατη τιμή για, για τη λιανική και τη χοντρική. Το περιθώριο που προτείνει η Κομισιόν είναι αρκετά γενναιόδωρο ώστε να επιτρέψει και νέε εισόδου, νέου ανταγωνιστέ στην αγορά. Αλλά η δική μα άποψη νομίζω ότι είναι ότι το παράκαναν λίγο, όπω είπα και κάποιοι ευρωβουλευτέ. Θα ήταν δυνατό να, υπάρχει, να υπάρχουν ανταγωνιστέ και με χαμηλότερα όρια και θα είχαμε και πάλι περιθώριο ανταγωνισμού. Υπάρχει όμω αρκετό περιθώριο στα ε, επίπεδα ανώτατων τιμών που υπάρχουν τώρα στο λιανεμπόριο και στο χοντρεπόριο. Μπορούν οι πάροχοι να μειώσουν τις τιμές τους και να καλύψουν πλήρω το κόστο του και να έχουν και κέρδο. Το μόνο που θα τους ε, υποκινήσει να το κάνουν αυτό είναι αν υπάρξει ένας νέος πάροχος στην αγορά, οπότε αυτό θα είναι αυτό που θα τους πιέσει για να μειώσουν τις τιμές. Πέντε λεπτά μου έχει δώσει ο πρόεδρος. Ε, ελπίζω να μπορέσω να σας απαντήσω. Αν δεν μπορέσω να σας απαντήσω τώρα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου, να μου στείλετε ένα μήνυμα κτλ. Ο πρόεδρος είπε κάτι για την ανάπτυξη των ε, πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Όντω, θα υπάρξουν τέτοιε υπηρεσίε, θα καταλήξουμε ε, σε πιο πανευρωπαϊκές ταρίφες, αλλά προς το παρόν αυτό δεν υπάρχει. Αλλά θεωρούμε ότι είναι δυνατό. Κύριε Κέφχαρτ, το ερώτημα για τα, για τα virtual structures δεν είναι ιονή λύση, είναι μια πραγματική λύση για να μειώσουμε την χρήση των υπηρεσιών δεδομένων και εντός της χώρας και στο εξωτερικό. Για να χρησιμοποιήσετε δηλαδή έναν πάροχο στο εξωτερικό με συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη τιμή για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Δεν θα είναι πολύ τεχνική η λύση αυτή, Δεν είναι εύκολο να γίνει. Δεν είναι δύσκολο. Ένα ερώτημα τώρα, ίσως φιλοσοφικό. Υπάρχει τελικά μια πραγματική αγορά και είναι δυνατή η ύπαρξη ανταγωνισμού. Ναι, θα πρέπει μάλλον να οριμάσει η αγορά κι άλλο, αλλά Σίγουρα ο στόχο μα θα πρέπει να είναι μια φυσιολογική ανταγωνιστική αγορά και ο ανταγωνισμό θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δυνατό να εξελιχθεί στο, σε μια τέτοια αγορά παρά τώρα. Ο κ. Ντεκάμπο είπε ότι όντω υπάρχουν τρει τρίτη πάροχοι που είναι έτοιμοι να μπουν στην αγορά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε μόνο στου εμπλεκόμενου φορεί. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν αυτέ οι νέε είσοδοι έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος, περισσότερο ανταγωνισμός. Ο πρόεδρος μου έδωσε 5 λεπτά, οπότε πρέπει να είμαι σύντομος. Λυπάμαι που σταματώ εδώ, αλλά ε, ευχαρίστω να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Ε, ξέρετε που είναι τα γραφεία μας. Είναι στη Ρήγα και θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε τα εγγένεια. Εάν θέλετε μπορείτε βεβαίως να έρθετε. Είσαστε καλοδεχόμενοι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω στα εγγένεια, αλλά δυστυχώ δεν θα μπορέσω να παραστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Λυπούμε που δεν μπόρεσα να σα ε, ε, να σας δώσω περισσότερο χρόνο, αλλά το πρόγραμμά μας είναι φορτωμένο όντως. Θα είμαστε βέβαια σε επαφή με την ΠΕΡΕΚ και η Κομισιόν άκουσε τα όσα είπε η ΠΕΡΕΚ σήμερα. Τώρα θα περιμένουμε την έκθεση της κυρίας Κόρχολα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε καταληκτικά σχόλια. Νομίζω καλύψαμε τα περισσότερα. Η κυρία Κόρχολα θα μας δώσει σε, κάποιο, σε κάποια μεταγενέστερη φάση και το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει. Η Επιτροπή Βιομηχανίας σήμερα το απόγευμα θα ορίσει και τον εισηγητή της, οπότε είμαστε πολύ μπροστά στο πρόγραμμα. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα για τον Κρίς Φοντέιν και τον ε, συνάδελφο του κύριο Νίμπλερ για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκανα σήμερα. Federica will look after you. I'm sorry I can't. going to keep that. I think he covered most of the points. Yeah. No, that's Federica's. Uh, yeah, I, I gave Federica back his Okay, ladies and gentlemen, can we... Um... και κύριοι, περνάμε σε ένα σημαντικότατο θέμα, νομοθετική πρόταση. Η οδηγία για πιστοτικές συμφωνίες σχετικές με κατοικία. Το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της, ε, της ε, βελτιωμένης συνεργασίας με άλλη ε, αρμόδια επιτροπή. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας θα φανούν και στην τελική μορφή του εγγράφου. Έχουμε τον κύριο Λέχνερ σαν εισηγητή ο οποίος ήταν εισηγητής και για τα θέματα της, της πίστοσης για τον καταναλωτή. Έχω και σκιώδεις εδώ αρκετές, αρκετούς, τον κύριο Φόξ και άλλους. Έχουμε επίσης και τον κύριο Πέλε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον καλωσορίσαμε προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο εκπρόσωπο της Προεδρίας προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Λέχνα να κάνει μια παρουσίαση σύντομη της έκθεσής του. Έχουμε 15 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας και να ζητήσω από τους υπολείπους να κάνουν σχόλια στην παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πω μόνο το πιο σημαντικά. Τις, ε, απλώς θα ε, υπογραμμίζω και κάποιες από τις παρατηρήσεις της γενικές που ήθελα να κάνω. Είναι αξιόλογη η πρόταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν βεβαίως έχει επιλέξει μια μετριοπαθή ε, έκθεση σε σχέση με παλαιότερες προτάσεις της που εντάξει μπορεί να μην καλύπτουν βέβαια τα πάντα. Εγώ ενσυνείδητα κρατήθηκα σε αυτό το πλαίσιο και θεωρώ ότι είναι σωστό και θα ζητήσω από τους ε, ε, συναδέλφους να μου πούνε εάν έχουν την ίδια άποψη. Ναι. Δεν έχω κάνει δηλαδή καμία διεύρυνση στο, θέμα. Υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά στην έκθεση, με την έκθεση Πρεσέντο που μιλούσε για προβληματικούς τομείς, για, άλλες, για, για κάποια άλλα προβλήματα τα οποία βεβαίως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια πράσινη βίβλο. Αλλά δεν ξέρω τώρα η Κομισιόν αν μπορεί να υποβάλει τέτοιες νέες ε, εκθέσεις χωρίς ε, μια αξιολόγηση επιπτώσεων, χωρίς μια κρόαση, χωρίς τίποτα, γιατί είναι και πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμα της ε, ΕΚΟΝ. Ο τίτλος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Δύσκολο να τον ε, διαχειριστούμε. Οι πράσινες, ε, οι πράσινες βίβλοι μιλούσαν για ε, δανεισμούς. Νομίζω ότι έπρεπε να βρούμε τελικά έναν καλύτερο τίτλο για την πρόταση και θεωρώ ότι είναι σημαντικό στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 ε, που συμπεριλάβαμε τις συγκεκριμένες αναφορές. Ένας ε, απλός αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να καταλάβει όταν διαβάζει για το πεδίο εφαρμογής ποια είναι τα βασικά σημεία. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για δάνεια για τις ε, κατοικίες, στεγαστικά δάνεια, αλλά για όλα τα είδη υποθηκευτικών τέτοιων δανείων έτσι ώστε ε, ο καταναλωτής να μπορεί να κατανοήσει. Αυτό προκύπτει και από το κείμενο που υπάρχει μέσα στο, στην έκθεση. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει σημαντική διαφορά και αυτό είναι ένα από του λόγου για το ότι είναι, μπορεί να είναι περιορισμένη η ολοκλήρωση τη αγορά. Μεταξύ των, του δικαίου για την ιδιοκτησία στα κράτη-μέλη μα υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει. Άλλο σημαίνει ε, δανειακή σύμβαση και υποθήκη στην, ε, στο Βρετανικό δίκαιο, άλλο στην, ε, ε, στις άλλες χώρες. Ας πούμε, η, στη Γερμανία όλοι παίρνουν α, υποθ, υποθηκευτικά δάνεια, τα οποία όμως δεν αποτελούν υποθήκη. Ουσιαστικά είναι μια δανειακή σύμβαση, αλλά σας λέω και πάλι ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. ας πούμε στην ε, Γερμανία ε, δεν είναι ε, τραβηγμένο από το μαλλιά να σας πω ότι μπορεί κάποιος να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσει μετοχές. Συμβαίνει αυτό. Όλα λοιπόν συμπεριλαμβάνονται και το, στην πρόταση και το θέμα είναι αν όντως πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τόσες πολλές λεπτομέρειες. Επίσης, ε, αν θα πρέπει άλλα είδη ε, δανειακών συμβάσεων να συμπεριλαμβάνονται. Πολλές φορές οι ε, η, όποιο θέλει να πάρει ένα δάνειο πούμε, για να ανοίξει μια επιχείρηση μπορεί να το κάνει μέσω ε, αυτή τη οδού. Να, χρησιμοποιήσει δηλαδή το, την ιδιότητα του ω καταναλωτή να πάρει ένα τέτοιο δάνειο και να μην το χρησιμοποιήσει όμω για το σκοπό που το πήρε, να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει μια ε, επιχείρηση. Και όταν ένα δάνειο εξαφαλίζεται μέσω μιας υποθήκης, ε, αυτό ε, ε, τότε ισχύει η οδηγία. όταν δεν καλύπτεται μέσω μιας υποθήκης δεν ισχύει η οδηγία. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και επίσης θα περιμένω να ακούσω τις απόψεις, να δω τα, τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ανώτερο όριο τα 2 εκατομμύρια επενδυτές ε, δεν νομίζω ότι χρειάζονται ε, την προστασία των απλών καταναλωτών. Και βεβαίω υπάρχουν και όλε οι, οι υπόλοιπες διατάξεις για το ίδιο κεφάλαιο. Ε, υπάρχουν πολλά, πολλά σημεία τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε και βεβαίω θα με ενδιαφέρε πολύ να ακούσω ποια είναι η άποψή σας. Νομίζω ότι αυτό το σημείο που αναφέρεται στα δύο εκατομμύρια θα πρέπει να ε, βγει από την οδηγία, να διαγραφεί. Επίσης, σε όλα τα σημεία όπου αναφέρω, ότι πρέπει να προβλέπονται, α, ή, να, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις για, τις, ε, για τα δάνεια, νομίζω ότι θα πρέπει να τις επεξεργαστούμε. Γιατί εδώ μιλούμε για την εξέταση των δανειακών συμβάσεων. Για, μιλούμε για διευκρινήσεις που μπορεί να χρειάζεται ένας καταναλωτής για να μπορέσει να συνάψει την δανειακή του σύμβαση. Να μην υπάρχει λοιπόν καμία ασάφεια. Θα πρέπει και στο κείμενο αυτό τα πράγματα να είναι απόλυτα σαφή. Στο σημείο 5 λέει ότι οι συνεργάτες των ε, τραπεζών θα πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή. Ε, ε εντάξει, αυτό ίσως να είναι λίγο μεταφραστικό θέμα, αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να μιλούμε για δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση του καταναλωτή και να έχουν, ε, ε, ο σκοπός τους να είναι να προστατεύσουν το συμφέρον του καταναλωτή. Όχι απλώς της τράπεζας. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το, το συμφέρον του καταναλωτή. Νομίζω ότι έτσι όπως ε, αναφέρεται είναι λίγο αποδυναμωμένο, λίγο ήπια η διατύπωσή του. Και το σημείο 8 επίσης πρέπει να αναδιατυπωθεί, γιατί ούτως ή άλλως κοστίζει αρκετά. Για τις διαφημίσεις επίσης δεν μπορώ να συμφωνήσω. Στις ε, βλέπω πολλές φορές ε, ε, αν θα, τι πρέπει να αγοράσω, από πού πρέπει να το αγοράσω, ε, πάει κανείς ας πούμε διακοπές και παντού βλέπει διαφημίσεις για υποθήκες, για δάνεια. Για δάνεια. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το α, περιορίσουμε. Άρθρο 9. Σημαντικό άρθρο. Πληροφορίες. Παροχή πληροφοριών πριν τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης τα φορολογικά ε, στοιχεία νομίζω ότι δεν ε, ε, πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ γιατί νομίζω ότι αποτελούν πρόσκομα προς την εσωτερική αγορά. Ένα ας πούμε υπάλληλο της μιας τράπεζας στην Πορτογαλία μπορεί ή θα πρέπει να ενημερώσει έναν Γερμανό ας πούμε πολίτη για το τι γίνεται με, την με τους φόρους που επιβάλλονται στην δανειακή του σύμβαση στη Γερμανία. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι και θέμα του καταναλωτή. Ο ίδιος θα πρέπει να ενημερωθεί και να φροντίσει για τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Προβλέπεται και στην οδηγία σχετική α, διάταξη για τις δανειακές ε, συμβάσεις, για την εξασφάλιση το, της χρηματοδότησης ότι ας πούμε το, το κεφάλαιο που έχει το, το, το, κεφάλαιο που θα πρέπει να έχει ο, ο, ο πολίτης που παίρνει το δάνειο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλό. Θέλω να πω απλώς ότι Εντάξει, μιλούμε για τις 14 ημέρες, για, για το περιθώριο που έχει να αποσυρθεί ο καταναλωτή, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός ή χρειάζεται άμεσα, τις, άμεσα το ποσό που θέλει να δανειστεί. Προφανώς ο καταναλωτή θέλει άμεσα, σύντομα, τα, το, τα χρήματα αυτά. Οπότε έχω κάποιες αμφιβολίες για αυτές τις συγκεκριμένε προθεσμίε. Νομίζω ότι αν πούμε απλώ άμεσα ή σύντομα θα έπρεπε να αρκεί. Η Κομισιόν ε, σε άλλα σημεία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση τη. Το άρθρο 9 όμω θα πρέπει να αποτελεί εναρμόνιση πλήρη και ε, ολοκληρωμένη. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, γιατί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προβλέπουν και επιπλέον πληροφόρηση. Γιατί η κατάσταση και ο κίνδυνος ε, με τη δύναμη του ε, σχετικού ε, του συμβατικού δικαίου μπορεί να είναι διαφορετική ένα περίπτωση, διαφορετική ένα περίπτωση. Οπότε να έχουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση μεν, αλλά ας μην αλλάξουμε τα πράγματα. Όταν ένα κράτος μέλος θέλει να είναι πιο διαφανές ας πούμε και θέλει να προβλέψει και άλλη πληροφόρηση, ή αν θέλει η τράπεζα η ίδια να δώσει επιπλέον πληροφορίες, θα πρέπει να προβλέπεται μέσα στην οδηγία να μπορεί να το πράξει. Άρθρο 11. Επαρκείς εξηγήσει. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, φορολογικοί συντελεστές, όταν είναι χαμηλοί, σε κάθε ε, περίπτωση, ακόμη και με μεταβλητούς ε, φορολογικούς συντελεστές, είναι εύκολο να αποπληρωθούν. Ε, οι μεταβλητοί είναι πολύ πιο, πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές από ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή που επιβάλλεται τελικά. Ίσως πολλές φορές ο καταναλωτής να, ε, να μην κατανοεί απόλυτα τι γίνεται με τα, ε, επιτόκια που ε, του επιβάλλονται. Σύμφωνα με τις ε, με τις διατάξεις που υπάρχουν μέχρι τώρα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικοί συντελεστές. Νομίζω ότι τουλάχιστον ο ελάχιστος Φορολογικό συντελεστή θα πρέπει να αναφέρεται. Ε, εντάξει, μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά όταν υπάρχουν ε, αναθεωρημένες, αναθεωρημένοι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι μπορεί τελικά να είναι πιο υψηλοί, ας πούμε για ένα δεκαετές δάνειο, θα πρέπει να δούμε πώς θα καθοριστούν. Άρθρο 14. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι, δεν, ότι μπορεί ο να υπάρξει άρνηση του ε, δανείου, τουλάχιστον έτσι όπως αναφέρεται εδώ στην πρόταση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, ας ε, πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ε, τεκμηρίωση. Ας πούμε για απαγόρευση δανειοδότησης κάποιου καταναλωτή. Κλείνοντας, να επανέλθω στο άρθρο 18 για την πρόορη εξόφληση και την αποζημίωση. Όταν ξέρει κανείς ότι αυτό είναι το πιο ακαθόδες θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τις διατυπώσεις αυτές ε, που, έχει, που έχουν επιλογή εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν, ε, υπάρχει πιθανότητα παρανόησης. Είχε κάποια στιγμή μπει η αποζημίωση και μετά κάποια στιγμή μπήκε μια δευτερεύουσα και διαγράφει τελικά ο όρος. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μην συμπεριλάβουμε οποιαδήποτε αλλαγή που κατά τα λοιπά βρίσκονται στο άρθρο 18. Να πω για τις πράξεις και το επίσης. Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν ε, απλώ κάνει μια σύντομη, υποβάλλει σύντομα την πρότασή τη και αν δεν περάσει, τότε έχει το δικαίωμα να την περάσει με την κατεξουδότηση πράξη. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό. Ε, η ε, της πράξης, δεν νομίζω ότι είναι α, αποδεκτές εδώ. Όταν κάτι δεν πάει καλά θα πρέπει και ο νομοθέτης, ε, η Κομισιόν, να μπορεί, να, ή το Κοινοβούλιο βεβαίως, να μπορεί να πει ότι μπορώ να ε, το αντιμετωπίσω με διαφάνεια, όχι μέσω των κατοξιότητας πράξεων. Και την, την περίοδο των δύο μηνών νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σύντομη. Για οποιοδήποτε περίπτωση, όχι μόνο για εδώ. Γιατί υπάρχουν ε, εκατοντάδε ε, κατεξοδότηση πράξη ε, κάθε χρόνο. Το Κοινοβούλιο σε δύο μήνε μπορεί ε, υποτίθεται να τις εξετάσει, αλλά μέχρι να τις δούμε όλες αυτές δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να γίνει σε δύο μήνες. Θα μπορούσαμε να πούμε τρεις, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε και πολύ περισσότερους να ζητήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν σχετικέ αλλαγέ. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. 26 Οκτωβρίου, 26 Οκτωβρίου, αν μπορεί να μου το επιβεβαιώσει και η γραμματεία, για, τις, για την υποβολή των τροπολογιών. Τέλος Νοεμβρίου ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή και ε, εμένα βασικά το ίδιο μου κάνει, αλλά για ένα τόσο σημαντικό θέμα Νομίζω ότι θα πρέπει να, να το προωθήσουμε άμεσα. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much for that comprehensive... Ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας. θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Οικονομική Επιτροπή. Ε, κάποιες από τις τροπολογίες τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ε, μελέτη ε, επιπτώσεων. Ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερος χρόνος. Λοιπόν, με τους κοιόδης τώρα. Πρώτος είναι ο κύριος Χουανγκόκ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Λέχνερ για την προσπάθειά του. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΚΟΝ ήταν κάτι δύσκολο και εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το συγκεκριμένο θέμα. Αξιολογώ θετικά επίσης και τον πραγματισμό που επέδειξε στα πλαίσια της δημιουργίας ενός διακανονιστικού πλαισίου σε μια αγορά η οποία δεν είναι ιδιαίτερα διεθνής και στην οποία αγορά μια περαιτέρω εναρμόνιση δεν είναι κάτι το οποίο ε, την χάνει προτεραιότητας. Δεν συμμερίζομαι όμως ε, τρία συγκεκριμένα θέματα τα οποία θέτει ο κ. Λέχνα. Και εδώ έχουμε μια ευκαιρία πρώτη συζήτηση. Το πρώτο θέμα αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του συστημικού κινδύνου. Σαν μέλος της Επιτροπής ΕΚΟΝ δεν νομίζω το ότι να περιοριστεί κανείς στους προσανατολισμούς της Επιτροπής της Βασιλείας είναι αυτού επαρκές. Ο συστημικός κίνδυνος των δανείων με υποθήκες είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί στην Ισπανία και την Ιρλανδία. Η Ένωση θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη στην πρόληψη αυτού του κινδύνου. Αυτό προστατεύει τον καταναλωτή αλλά είναι και θέμα γενικότερα οικονομικής σταθερότητας. Διαρωτώ με για την εξαίρεση από την οδηγία των πιστώσεων που δίδονται στους εργολάβους. Αυτό είναι ένα θέμα που θέσατε προηγουμένως, στους κατασκευαστές καλύτερα. Διότι οι κατασκευαστές είναι στόχος του ανωτάτου ορίου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως οι κανόνες θα πρέπει να προσαρμεστούν σε κάποιες τοπικές προτεραιότητες, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση φοβάμαι ότι ε, κάνουμε ένα σημαντικό λάθος σε σχέση με την οδηγία. Τρίτον, παρά την ύπαρξη κανόνων που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, ε, δεν είμαι σίγουρος για την ευθυγράμμιση της οδηγίας αυτής με την οδηγία ε, για την καταναλωτική πίστη. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί, το θέμα που μας απασχολεί απαιτεί εξειδικευμένες απαντήσεις πέραν των, των υπαρχουσών ρυθμίσεων. Και νομίζω ότι το περιθώριο που δίνουμε στα κράτη-μέλη εν μέρη λύνει το πρόβλημα. Και τέλος, και εδώ είναι διαφορετικό το θέμα, διαρωτώμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των λεγόμενων βοηθητικών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά και ε, Κατά τη διάρκεια της συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να το εμβαθύνουμε. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much indeed, Mr. Uh, Mr. Bozoi is next. Thank you very much, Chairman. Uh, I would like to congratulate her. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την προσπάθεια που έκανε να ετοιμάσει την πρόταση αυτή για τα ανεπόθηκα ε, δάνεια. Φυσικά και υπάρχουν ε, πολλές καλές προτάσεις που θα υποστηρίξω τώρα για το συνολικό κόστος του δανείου. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους ε, καταναλωτικής πίστης. Συμφωνώ ότι, όταν, ότι το κόστος δεν θα πρέπει να, το κόστος της δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συνολικού κόστους. Υπάρχει κάποιο κόστος το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει αυτός που παίρνει το δάνειο, όπως ε, για την εγγύηση όσον αφορά το κτίριο, όταν ε, πρόκειται για ανυπόθηκο κλπ. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να διαλέξει το συμβολογράφο για παράδειγμα, οπότε να ξέρει κάθε φορά ποιο θα είναι το κόστος που θα πέσει στους ώμους του. Στο σημείο 12 που αναφέρεται το ποσοστό και το συνολικό κόστος, πρέπει να το ξαναδούμε. Βέβαια, ως ε, αυτός που δανείστε πρέπει να ενημερωθεί από τον πιστωτή για το κόστος και των υπηρεσιών του πιστωτή. Αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στις διαφημίσεις. Νομίζω ότι τόσα λέει για την διαφήμιση η Κομισιόν είναι υπερβολικά γιατί τελικά θα είναι αδύνατο να κάνει διαφήμιση ο πιστωτής στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, γιατί εκεί είναι πολύ σύντομες οι διαφημίσεις. Ενώ αν συμπεριληφθούν όλες αυτές οι πληροφορίες που λέει η Επιτροπή θα γίνει ανέφικτο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για το συνολικό κόστος που επομίζεται ο καταναλωτής και να ξέρει ότι θα χάσει την ιδιοκτησία του αν δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Όπως λέει και ο κύριος Λέχνερ, έτσι και εγώ πιστεύω ότι τους κινδύνους αυτούς τους ξέρει όταν βάζει ένα υπόθηκο δάνειο ο καταναλωτής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι πληροφορίες είναι πληροφορίες που θα έπρεπε να παίρνει ο καταναλωτής στο προσυμβατικό στάδιο. Νομίζω ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία πρέπει να αποφασίσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όχι η Κομισιόν. Οπότε συμφωνώ με τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις συμβατικές πληροφορίες τώρα, νομίζω ότι προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία για όλα τα πιστοτικά ιδρύματα και τους ενδιάμεσους, ώστε να υπάρχει επίσης και η ίδια προστασία για όλους τους καταναλωτές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήσιμο θα ήταν να έχουμε μια όσο γίνεται μεγαλύτερη εναρμόνιση. Για τις κατεξουδότητες πράξεις τώρα, συμφωνώ με την προσέγγιση του κυρίου Λέχνερ, περιορίζοντας το εύρος τους. Και το τελευταίο μου έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια αρνητική αξιολόγηση κατά καταναλωτή, δεν θα έπρεπε ο πιστωτής να δίνει δάνειο. Εδώ πρέπει να βρούμε ένα, μια μέση οδό και συμφωνώ να πάμε προς το δρόμο που προτείνει ο κύριος Λέχνερ. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να φαίνεται, από την... να φαίνεται ότι έχει γίνει πραγματικά αξιολόγηση του καταναλωτή. Στην περίπτωση πάντως που αρνηθεί ένα πιστοτικό ίδρυμα το δάνειο, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε όλα τα στάδια βάσει των οποίων οδηγήθηκε σε άρνηση στον καταναλωτή ο πιστοτής δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους στόχους της οδηγίας. Εννοείται ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για τη βάση δεδομένων και για το δικαίωμά τους να αλλάζουν κάθε μήνα την απόφασή τους. Αλλά ο πιστωτής δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει κάθε φορά. Κατά τη γνώμη μου φωτώνουμε υπερβολικά το σύστημα έτσι. Αυτά είναι κάποια μόνο θέματα που ήθελα να σας αναφέρω. Υπάρχουν και άλλα που έχω υπόψη μου και από αυτόν θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαρίστως να συνεχίσουμε τη ζήτηση για όλα αυτά τα θέματα με τους άλλους κοιόδες και με τον εισηγητή στο μέλλον. Ευχαριστούμε η κυρία Ρίλελ και μετά ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα γιατί συνεργαστήκαμε και όσον αφορά την οδηγία για την προστασία του καταναλωτή. Είναι σωστή η προσέγγιση του. Όταν συζητήσαμε για τα ανυπόθηκα δάνεια τότε, είχαμε πει ότι δεν θέλουμε έμεσα να είναι ανοιχτή η αγορά. Θέλουμε να υπάρχει προστασία στον καταναλωτή. Και ο κύριος Λέχνερ ε, το τήρησε. Οι προτάσεις του βρίσκω ότι είναι λογικές και σωστές. Έλαβε υπόψη του αυτά τα οποία είπαμε και για την ε, καταναλωτική πίστη. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα ώστε να μην υπάρχουν ασυνέπειες. Όσοι δουλεύουν στον τομέα της καταναλωτικής πίστης δεν το γνωρίζουν πάντα. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχουν παρόμοιες ρυθμίσεις και στις δύο περιπτώσεις. Για το θέμα του χρονοδιαγράμματος τώρα, εγώ προσωπικά Συμφωνώ με τον κύριο Λέχνερ ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Οικονομική Επιτροπή για να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν ε, υπάρχει ικανοποίηση από όλε τις ε, πλευρές για την έκθεση της ε, Οικονομικής Επιτροπής. Γι' αυτό και επιμένω ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας. Πρέπει να τα συζητήσουμε ακόμα και να πιέσουμε την Επιτροπή ΕΚΟΝ ώστε η συζήτηση να είναι ευρύτερη. Δεν βλέπω γιατί μας πιέζουν τόσο πολύ. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα καλό είναι να μας δοθεί ευκαιρία να δουλέψουμε σωστά, γιατί οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι τεράστιες αν πάρουμε λάθος αποφάσεις. Τέλος, για μένα η κατεξοδότηση πράξης είναι κάτι για το οποίο συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λέχνερ. Σε όποιο τομέα και αν δουλεύουμε, είτε πρόκειται για ρύθμιση για τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα, το ίδιο πιστεύω ότι η Κομισιόν πρέπει να ετοιμάζει καλύτερα τις προτάσεις της για να έχουμε λιγότερες κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ευχαριστώ. Mr. Fox. Uh, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λέχναρ για τη δουλειά του και για την πραγματιστική του στάση και σε σχέση με αυτόν που δανείζεται και σε σχέση με αυτόν που δανείζει. Όπως είπα έχω πολλές επιφυλάξεις για τις προτάσεις της Επιτροπής και γι' αυτό υποστηρίζω την τροπολογία 79 που απαιτεί από την τράπεζα αν οι συμβουλές που δίδονται βασίζονται μόνο στα δικά τους προγράμματα και, παράγω, και προϊόντα και όχι από την υπόλοιπη αγορά συνολικά όπως θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιλαμβάνει θα έλεγα και κάποια περιφερειακά προγράμματα τα οποία ρυθμίζονται καλύτερα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν τον, τον καταναλωτή και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, να δημιουργήσουμε προβλήματα, να αλλάξουμε ε, τις ρυθμίσεις. Ε, πρέπει να εξαιρέσουμε λοιπόν από το της οδηγίας κάποιους ε, μορφές δανεισμού όπως τον λεγόμενο κοινωνικό δανεισμό και κάποιες επίσης ενυπόθηκες μορφές δανεισμού δεν είναι κατάλληλες όπως ε, οι επενδυτικές αγορές από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και τα λεγόμενα δάνεια γέφυρες ή ενδιάμεσα δάνεια. Δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές τις περιπτώσεις οι ρυθμίσεις που προτείνονται. Σημερίζομαι λοιπόν τις ανησυχίες του εισηγητή σε σχέση με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, να ακούσει αυτά τα οποία λέμε. Συμφωνώ με ένα δελτίο ευρωπαϊκό το ίσες ενημέρωσης. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ένα τέτοιο μέτρο με υψηλό κόστος. Θα ήθελα λοιπόν ε, να υπάρξει επιλογή ανάμεσα στο ίσες ή ένα αντίστοιχο εθνικό έγγραφο το οποίο έχει εγκριθεί όπως είπα από τον εθνικό ρυθμιστή και περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες. Όπου υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει λόγος να το κρεμίσουμε και να χτίσουμε ένα καινούριο. Επίσης η τροπολογία που υποχρεώνει ε, τις τράπεζες να δίνουν εξηγήσει για αρνητική απάντηση σε αίτηση δανειοδότησης ε, και επίσης οι ρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι σωστές. Ε, μια αξιολόγηση αρνητική για κάποιους σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει δάνειο, αλλά δεν θα ε, υπάρξει δυνατότητα για καμιά καλύτερη ευελιξία και η ελευθερία σύμβασης ανήκει τελικά στους εταίρους και αυτοί αποφασίζουν αν θα δώσουν συνέχεια ή όχι στην αίτηση σχετικά με την ανάγκη στοιχείων η αναζήτηση και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι πάρα πολλές πληροφορίες δεν βελτιώνουν ε, τη στάση του καταναλωτή. Δεν πρέπει να πνίξουμε τον καταναλωτή με πάρα πολλές πληροφορίες. Οι υποθήκες δεν πολλούνται επί τη βάση μιας απλής διαφήμισης και γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε σε επίπεδο ενημέρωσης, σε λίγες αλλά βασικές αρχές ενημέρωσης. Και τέλος, ο κύριος Λέχνερ εισάγει ένα μέτρο το οποίο ζητάει μια γρήγορη επιστροφή που συμπεριλαμβάνει την απώλεια του κόστους των επιτοκίων, ενώ εμείς θα θέλαμε να κρατήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν επιβαρύνει τόσο τον καταναλωτή. Τέλος, Πρόεδρε, είναι απαραίτητο να μην πάρουμε μέτρα τα οποία να δεσμεύσουν ακόμα περισσότερο την παροχή δανείων και πίστοσης σε μια τόσο δύσκολη περιοχή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνει προτάσεις αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσει. Ευχαριστώ τον κύριο Λέχνερ και τους άλλους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Μας είπατε πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τα σχόλιά σας είχαν ενδιαφέρον και είμαστε ακόμα στην αρχή. Ε, κάποια άλλα μέλη θα ήθελαν το λόγο, η κυρία Βάιλερ πρώτα. Και μετά θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσει το θέμα πριν περάσω πάλι στον κύριο Λέχνερ μάλλον να το κλείσει. Βάιλα κάποια ερωτήματα, γιατί δεν είμαι και ειδική. Έχω κάποια προβληματάκια με την επιχειρηματολογία που έχουμε εδώ συμπεριλάβει. Ότι, για παράδειγμα, η διαφήμιση δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για, τους, για όσους κάνουν αίτηση για δάνειο. Ίσως εγώ να μην έχω καταλάβει καλά, αλλά το έχουμε ίσως να, πρόκειται και από άλλες οδηγίες ή από άλλα κείμενα. Απλώς θέλω να εξασφαλίσουμε ότι οι ετούντε ε, όσο όποιος αιτείται να πάρει δάνειο, μπορεί να ε, ενημερωθεί, εν πάση περιπτώσει, αν όχι από την διαφήμιση, από κάπου αλλού. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται και για τις ασφαλιστικές, ε, για τα ασφάλειες που συνάπτουμε Ωραία, να μην είναι η διαφήμιση το σωστό μέσο, αλλά εν πάση περιπτώσει από κάπου πρέπει να ενημερωθεί ο δανειολήπτη. Ε, επίσης, οι κακέ εμπειρίε που έχουμε τα τελευταία δέκα χρόνια που έχουμε δει και μέσω της ε, εμπειρία μα από την Ισπανία, αυτά μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε. Υπάρχουν κάποια διδάγματα που να έχει εξάγει η Κομισιόν από όλη την ε, ιστορία αυτή, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις από το να ξανασυμβούν στο παρελθόν. Στο μέλλον, συγγνώμη. Α κάνουμε λοιπόν με τη νέα νομοθεσία ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε. Και ένα τελευταίο σημείο, ε, θέλω να σα συγχαρώ κύριε Λέχνερ, γιατί τα δικαιώματα που έχει εδώ το Κοινοβούλιο νομίζω ότι θίγονται επαρκώς στην έκθεσή σας και όντως ε, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και θα έχετε βεβαίω και την στήριξή μα στην νομοθεσία σα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε τα σχόλια της Κομισιόν. Όπως είπε και η κυρία Βάιλερ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των κατεξιοδότηση πράξεων και τις οποίες, πολλές από τις οποίες έχουμε απορρίψει εμείς μέσω των δικών μας διαδικασιών για τον λόγο ακριβώς του υψηλού αριθμού που λαμβάνουμε. Αν μπορείτε σε πέντε λεπτά να μας απαντήσετε, έτσι ώστε να έχει και ο εισηγητής τον λόγο για να απαντήσει. Ο κύριος Πέλε, ευχαριστώ πολύ. Γαλλικά θα μιλήσω αυτή τη φορά. Πεντέμιση σημεία έχω. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τις πληροφορίες και τις επεξηγήσεις τους. Η Επιτροπή εννοείται ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Πρώτον, η Κομισιόν σημειώνει ότι υπάρχουν διάφορες τροπολογίες στο σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Λέχνερ που θέλουν να ευθυγραμμίσουν τις διατάξεις της πρότασής μας με τις διατάξεις της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η πρόταση σχετική με τα ενυπόθηκα δάνεια ακολουθεί τη δομή της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, ιδιαίτερα όσον αφορά την πλαισίωση της διαφήμισης με έναν κατάλογο πληροφοριών που πρέπει να δίνονται, όσον αφορά επίσης το τυποποιημένο δελτίο και τις επεξηγήσεις που πρέπει να δίνονται για την καλή κατανόηση του προϊόντος και τη συγκρισιμότητα και όσον αφορά τη χρησιμότητα του δανειολήπτη, ε, του δανειδότη, συγγνώμη, να κρίνει την εξοπιστία του δανειολήπτη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Έπειτα οι όροι και ορισμοί κλειδί που ε, χρησιμοποιούνται για την καταναλωτική πίστη συμπεριλαμβάνονται και στην τρέχουσα πρόταση. Συγχρόνως νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η ιδιαιτερότητα των ενυπόθηκων δανείων που δίνονται για την απόκτηση κατοικία. Και ακριβώ επειδή υπάρχει εδώ ιδιαιτερότητα, γι' αυτό έχουμε και μια κάπω διαφορετική προσέγγιση. Φυσικά και παίρνουμε μαθήματα από την οικονομική κρίση. Και έτσι φροντίζουμε τα δάνεια να δίνονται εφόσον υπάρχει υγιής βάση. Γι' αυτό και οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του δανειολήπτη είναι πιο αυστηρά από ό,τι ήταν στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Επίσης, οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με το τυποποιημένο δελτίο, σε ποια στιγμή πρέπει να δίνεται αυτό, εδώ είμαστε πιο συγκεκριμένοι από ότι είμαστε για την καταναλωτική πίστη. Το μισό μου τώρα σημείο έχει να κάνει με το ότι κάποιες τροπολογίες απορρέουν νομίζω από προβλήματα μετάφρασης στα γερμανικά, εκεί όπου δεν υπάρχει διαφορά ε, τη, ανάμεσα στην καταναλωτική πίστη και την ενυπόθηκη. Αυτό είναι θέμα των γλωσσολόγων να το βρουν, των γλωσσικών ειδικών. Τέλος, ε, προτείνονται διάφορα πράγματα στις τροπολογίες 25 με 33, πράγματα τα οποία δεν έχουμε συμπεριλάβει. Και δεν τα έχουμε συμπεριλάβει επειδή δεν έχουμε καμία απόδειξη για την αναγκαιότητά τους. Να σας υπενθυμίσω, ναι, με 33 αναφέρονται στις, ε, αποκλείει το CSD. Τέλος. Το άρθρο το σχετικό με τις προσεβατικές πληροφορίες. Εδώ θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ε, πρότασή μας. Άλλο είναι οι γενικές πληροφορίες και άλλο είναι οι εξατομικευμένες πληροφορίες. Το άρθρο 9.1 της πρότασης συμπεριλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες προς το καταναλωτή ανά πάσα στιγμή για όλα τα προϊόντα που προσφέρει ο δανειοδότης. Εδώ έχουμε επίσης και την ιδέα του κώδικα δεντολογίας που είχε εγκρίνει σε σύστασή της το Μάρτιο του 2001 η Επιτροπή. Ο κατάλογος όμως των στοιχείων που δίνονται εδώ δεν πρέπει να ευθυγραμμιστεί στις τυποποιημένες πληροφορίες που δίνονται βάσει του τυποποιημένου δελτίου το άρθρο 9.2 της πρότασης. Αυτό αναφέρει την ιδέα μιας προσεβατικής τυποποιημένης ε, ενός δελτίου τέτοιου. Δεν υπάρχει κατάλογος πληροφοριών, δηλαδή στο σώμα της οδηγίας, σε αντίθεση με το όσο είχαμε για την καταναλωτική πίστη, δεδομένου ότι εδώ πέρα τα ανυπόθηκα δάνεια είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τέταρτο σημείο μου. Και ο κύριος Λέχνερ το ανέφερε ο συγητής, αλλά και κάποιοι σκιώδεις. Πρόκειται για το βαθμό εναρμόνισης της οδηγίας. Η τροπολογία 90 ζητάει ανώτατη εναρμόνιση. Είναι αλήθεια, γιατί όχι στο κάτω-κάτω. Αλλά εμεί δεν πιστεύουμε ότι μια πλήρης εναρμόνιση είναι ε, αναγκαία ή κατάλληλη, γιατί η δομή των ενυπόθηκων ε, δανείων διαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και τα προϊόντα χρηματοδότησης κάτι το οποίο υπογραμμίσατε κι εσείς. Η ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον είναι καλά στοχοθετημένη και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η πρόταση οδηγίας πρέπει να αφήνει ένα περιθώριο ελιγμών αρκετά μεγάλο στα κράτη-μέλη εφόσον αυτό δικαιολογείται. Αυτό πιστεύουμε και εμείς όταν πρόκειται για την, ε, ε την επιστροφή των χρημάτων νωρίτερα από το συμφωνημένο. ενώ από την άλλη η τυποποιημένη ε, προσυμβατική ενημέρωση πρέπει να είναι εναρμονισμένη. Το τελευταίο μου σημείο προς το παρόν έχει να κάνει με το εξή. Το προσχέδιο ζητά την κατάρριξη διάφορων κατεξουσιοδότηση πράξεων. Υπάρχει η τροπολογία 49 φυσικά, που η 50 για τη διαφήμιση, 61 για τις πληροφορίες που δίνουν οι μεσίτες, η 66 για τους υποθέμενους υπολογισμούς, η 77 για τη βάση δεδομένων, η 80 επίσης κλπ. κλπ. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έκανε την πρότασή της και εισήγαγε όλες ε, αυτές τις κατεξουδότηση ε, πράξεις δεν ήταν για να το κάνει σε βάρος του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου αλλά για να προσαρμοστεί στις εξελίξεις στην αγορά. Υπάρχουν νέα προϊόντα στην αγορά ή επειδή υπάρχουν νέες πρακτικές στην αγορά. Για τον υπολογισμό του ΤΙΑΖΕ, για παράδειγμα. Όπως και να έχει πάντα το πράγμα. Εφόσον οι σε αυτές πράξεις πρέπει να καταργηθούν, να βγουν δηλαδή από την πρόταση, τότε θα πρέπει να βάλουμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Για παράδειγμα το ποσό της ε, ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Είμαστε σήμερα σε θέση να τα κάνουμε όλα αυτά ή μήπως πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να τα μελετήσουμε, αλλά η πρόταση έχει τη δικιά της αξία και τη χρησιμότητα. Βάσει της Επιτροπής λοιπόν η πρόταση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον όγκο των υπόθηκων δανείων που δίνονται γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλά ζυγισμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις ξεκάθαρες απαντήσεις που μας δώσατε. Συνεπώς, ο κύριος Λέχνε τώρα για να συνοψίσει. Παρακαλώ. Και να μας υπενθυμίσει το χρονοδιάγραμμα, το προσωρινό τουλάχιστον. Χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις με την Οικονομική Επιτροπή, έτσι, για να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν, να ευχαριστήσω και τους συνάδελφους για την παρέμβασή τους. Θα εξετάσω βεβαίως, θα σκεφτώ όλα όσα είπατε. Νομίζω όμως ότι η πρότασή μου γενικώ έτυχε έτσι θετικής αποδοχής από, τις, από τους συναδέλφους. Χαίρομαι όμως που θα συμπεριλάβουμε και τις συζητήσεις ε, με την ΕΚΟΝ. Προφανώς μεταξύ των καταναλωτικών δανείων και των ε, στεκαστικών δανείων υπάρχει διαφορά, αλλά αν τώρα αυτό έχει να κάνει με την, ε, με την πίστη του δανειολήπτη ή όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το, να, το, να το καταδείξουμε στην διατύπωση του κειμένου. Νομίζω ότι αυτό που λέει αρκεί ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή. Γιατί η οδηγία για την καταναλωτική πίστη είναι και υποχρεωτική. Ε, τα κρατημέλη δηλαδή θα πρέπει να κάνουν τι. Αυτή τη στιγμή να διατηρήσουν ένα, δύο διαφορετικά ε, ε συστήματα ή να υποχρεώσουν τους καταναλωτές τους να υπόκεινται σε δύο διαφορετικές διατάξεις. Ε, για την κυρία Βάιλερ. Ε, όντως, κανένας δεν ε, περιμένει να είναι όλα πάρα πολύ ωραία και πολύ θετικά και πολύ αισιόδοξα από τις ε, ε, διαφημίσεις. Ε, προφανώς και δεν χρειάζεται υπερπληροφόρηση των καταναλωτών, αλλά στο άρθρο 9 πρέπει να εξασφαλίσουμε ποιες είναι οι πληροφορίες που θα δίνονται στον καταναλωτή. Βεβαίω αυτό δεν αναφέρεται στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη, παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αντίφαση εδώ μεταξύ των δύο. Υπάρχουν πρότυπες, υπάρχουν στάνταρ, τυποποιημένες πληροφορίες που λαμβάνει ο, α, ο καταναλωτής και νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να τις έχει. Επίσης θα πρέπει να έχει και χρόνο για να τις μελετήσει αυτές τις α, πληροφορίες που του δίνονται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημεία, από τις λεπτομέρειες ίσως, που είναι, σημαντικό, που είναι σημαντικές για τα κράτη-μέλη. Να μπορούν δηλαδή και αυτά να μελετούν την αξιοπιστία του κάθε καταναλωτή πριν δώσουν το δάνειο. Τώρα για το άρθρο 8 που είπε ο κύριος Φόξ. Α, δεν είναι εδώ ο κύριος Φόξ. Α, έφυγε ο κύριος Φόξ. Μάλλον δεν κατάλαβε καλά το άρθρο 8 ο, ο, ο κύριος Φόξ. Η Κομισιόν κάτι διαφορετικό λέει από αυτό που κατάλαβε ο κύριος, ε, ο κύριος Φόξ. Δεν μιλούμε δηλαδή για, ε, για, ζημιά, για αποζημίωση, μιλάμε για ζημιά. Εγώ θα Ξανασυζητήσω με τον συνάδελφο Πρεσέντο, το έκανα και σήμερα. Πήγαν πολύ καλά οι συζητήσει. Θα δούμε πώ θα προχωρήσει η όλη διαδικασία με τι διαπραγματεύσει. Χαίρομαι όμω για την αποδοχή που δείξατε στην έκθεσή μου και υποθέτω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια πολύ καλή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Χαίρομαι που έχουμε προχωρήσει σε αυτό το σημαντικό θέμα. Ξέρετε ο κύριος Λέχνερ θα μας διαφωτίσει και θα μας ενημερώσει και για το χρονοδιάγραμμα και όλα τα θέματα τα οποία μείνε σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, τελευταία έκθεση είναι η γνωμοδότηση την οποία προετοιμάζουμε για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την οδηγία για τις επιτρεπόμενες χρήσεις των λεγόμενων σε εισαγωγικά ορφανών έργων. Έχουμε τον εισηγητή και τις σκιώδεις εισηγήτριες Πέντεργαστ, Ρόιτεβα. Κύριος Φόξ έφυγε, ίσως να ξανάρθει όμως. Χαίρομαι επίσης γιατί καλωσορίζω τον Διευθυντή της Αρμόδιας ε, υπο... Ε, ε, διεύθυνσης της Επιτροπής, τον κύριο Μάνφρετ Φρόιλιγκα ο οποίος είναι γνωστός φίλος της Επιτροπής μας. Θα απαντήσει λοιπόν και αυτή όταν είναι εδώ. Μάγδα, σε καλωσορίζουμε. Λοιπόν, κύριε Μάντερς, μπορείτε να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ την Μπάρμπρα γιατί είναι τα γενέθλιά της. Καμία σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, αλλά φυσικά χρόνια πολλά. Και ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, καμία σχέση με τα, με τα έργα αυτά. Λοιπόν, λίγα λόγια για την πρόταση αυτή. Τι είναι τα ορφανά έργα λοιπόν είναι έργα των οποίων ε, οι κάτοχοι δεν μπορούν να εντοπιστούν και να ευρεθούν. Και όταν ένα έργο διατίθεται στο κοινό, τίθεται το θέμα της εφαρμογής των αρχών της, ε, ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά δεν υπάρχει, οπότε είναι ένα πρόβλημα. Η οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις ε, για την ε, συντήρηση προϊόντων, αλλά δεν δίνουν την δυνατότητα στις βιβλιοθήκες σαν παράδειγμα να καταστήσουν ε, το υλικό αυτό διαθέσιμο ψηφιακά ακόμα και για μη εμπορικούς λόγους. Και η πρόταση η οποία γίνεται δίνει την δυνατότητα νομικής ασφάλειας για να περάσουν σε αυτό το στάδιο οι βιβλιοθήκες. Λόγω του ότι υπάρχει ένα κοινό λοιπόν στην συγκεκριμένη οδηγία και δημιουργείται στρέβλωση πιθανώς στην εσωτερική αγορά, με την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε αρχεία, σε σχολεία, σε βιβλιοθήκες να παρέχουν τα έργα αυτά online στον ψηφιακό κόσμο όπως γίνεται τα ορφανά αυτά έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε ε, την διαδικασία αμοιβαία αναγνώρισης εθνικών λύσεων γιατί ορισμένες χώρες έχουν τέτοιου είδους λύσεις. Δύο-τρεις χώρες ήδη εργάζονται με την συγκεκριμένη δυνατότητα αναγνώρισης των ορφανών έργων και πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και είναι καλή η ιδέα της αμοιβαία αναγνώρισης και ελπίζω να περάσει πιο εύκολα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια σημαντική αναφορά στη ρύθμιση για τη βιβλιοθήκη Google στις Ηνωμένε Πολιτείε, την ψηφιακή βιβλιοθήκη Google. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ του πώς ένα τέτοιο θέμα μπορεί να επιληθεί με ικανοποιητικό τρόπο για το μέλλον ακόμα και για αυτούς που έχουν την πνευματική ιδιοκτησία. Είναι καλή η πρόταση. Κατέθεσα πολλές τροπολογίες. Ε, ε, Κατέθεσα πολλές τροπολογίες γιατί πιστεύω ότι ακόμα και μια καλή πρόταση μπορεί να βελτιωθεί. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τον συγκεκριμένο ρόλο που έχει η πνευματική ιδιοκτησία. 15 είναι οι τροπολογίες. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο αφορά θα έλεγα μια πολύ δημιουργική και εφάνταστη δραστηριότητα, αν και κάποιοι συνάδελφοι ίσως να διαφωνήσουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η ανάγκη να υπάρξουν τα μέσα για την προστασία της πνευματικής κληρονομιάς και γι' αυτό κατέθεσα την τροπολογία 1. Εάν και όταν ο κάτοχος του δικαιώματος εμφανίζεται, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει έρευνα στα κράτη-μέλη, να δούμε πού δημοσιεύθηκε το έργο πρώτο, που γνωστοποιήθηκε στο κοινό και γι' αυτό προτείνω λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή κάποιες τροπολογίες. Η έρευνα θα πρέπει να γίνει με λογικό τρόπο και καλή την πίστη, διατηρώντας πάντα σε πρώτη θέση το δημόσιο συμφέρον. Αν δημοσιευθεί ήδη το έργο σε άνω του ενός κράτους μέλους ταυτόχρονα, αυτό είναι κάτι το εφικτό και απαιτείται να υπάρξει μια λύση. Then the right holders, uh, amendment. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων, τώρα 12 με 14 οι τροπολογίες αυτές. Όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους πρέπει να έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Και όχι μόνο στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη όπου δημοσιεύτηκε το έργο για πρώτη φορά, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. και θα πρέπει να αμυφθούν γι' αυτό όταν δημοσιεύεται το έργο. Η βάση δεδομένων την οποία χρειαζόμαστε στην Ευρώπη θα πρέπει, βάσεις δεδομένων που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές έτσι ώστε να είναι εύκολο να ψάξει κανείς να βρει το ποιος είναι ο πνευματικός εισαγωγικά ιδιοκτήτης. Προσθέτω ότι η οδηγία αυτή πρέπει να αφορά υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ρυθμίσεις. Η νομοθεσία πρέπει να ισχύει και στο μέλλον. τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίζουν σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία ρυθμίσεις όπως οι λεγόμενες συλλογικέ ε, άδειε. Εν πάση περιπτώσει αυτά λέγουν οι τροπολογίες και περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων να μου πούν αν έχουν κάτι να προτείνουν στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ οι συνάδελφοι. Κυρία Ρόιτεβα. Ευχαριστώ. Στηρίζω απόλυτα το σχέδιο αυτό και χαίρομαι που το ετοίμασε η Επιτροπή. Θέλω όντω να προχωρήσει γρήγορα και απρόσκοπα η πρόταση αυτή. Είναι σημαντικό η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη στην Ευρώπη να είναι συμβατή με το Google, το οποίο βρίσκεται πολύ μπροστά. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε 200.000 ταινίες, πάρα πολλές φωτογραφίες και ξέρω πόσα βιβλία, πάρα πολλά. Ένα πράγμα μου λείπει εμένα από αυτή την πρόταση. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να έρθω λιγάκι και στην τελευταία τροπολογία του εισηγητή, στο άρθρο 3 δηλαδή, ή μάλλον όχι, είναι το άρθρο 7, σημείο 5α. Λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη για να πληρώσουν. Όμως τελικά οι βιβλιοθήκες είναι αυτές που θα πάρουν το έργο, οπότε πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε και γλωσσικά να υπάρχει πρόσβαση. Δηλαδή, οι τίτλοι και τα ονόματα να προσφέρονται ε, με μεταφράσεις στη κάθε εθνική βάση δεδομένων για να μπορούμε πιο εύκολα να τα βρούμε. Αλλά ξεκινήσουμε βέβαια από το να βρούμε τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Πάντως ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα, ένα κεντρικό δίκτυο ή να υπάρχει διασύνδεση αν μη τι άλλο με όλες τις άλλες χώρες. Τι θα γίνει αργότερα στο μέλλον. Δεν θα πρέπει κάθε φορά να ασχολούμαστε με την διαλουργικότητα 27 διαφορετικών συστημάτων και να αρχίζουμε κάθε φορά από την αρχή. Ας φροντίσουμε λοιπόν αν μη τι άλλο να υπάρχει ένα σύστημα. Έπειτα θα υπάρξει ένας μεγάλος κατάλογος οργανισμών ώστε να μπορεί να γίνει η ψηφιοποίηση και από άλλες οργανώσεις και να συμπεριλάβουμε και όλα τα έργα τέχνης. Ίσως λοιπόν πρέπει να επεκτείνουμε την πρόταση αυτή και σε μαγνητοσκοπήσεις και σε φωτογραφίες και σε έργα τέχνης. Ξέρω ότι θα είναι περίπλοκο και δεν θέλω να καθυστερήσουμε με την έγκριση της ρύθμισης αυτής. Να κοιτάξουμε όμως λιγάκι τι γίνεται και με τις αλλαγές στα σύνορα που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο αιώνα ή αυτόν, για να μην εισμάτι κάνουμε προσπάθειες. Συμφωνώ εδώ με τον εισηγητή. Έπειτα από πού ξεκίνησαν τα έργα τέχνης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να λυθεί με την πρόταση αυτή. Όμως μπορεί να έχουν εμφανιστεί στο κοινό σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, λέμε ότι το 30% των βιβλίων τυπώθηκαν στην Ινδία. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 6. Εδώ δεν νομίζω ότι πρέπει να περιορίσουμε το δικαίωμα στην χρήση ε, πλήρων καταλόγων. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εγκυρότητα κάθε φορά που ζητάμε από τις βιβλιοθήκες να πληρώσουν για την χρήση έργων τέχνης. Πρέπει να υπάρχει πραγματικά κάτι που να στέκει νομικά. Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο. πρέπει να συμμετέχουμε και στην συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο για αυτό το θέμα και να δούμε τι λέει το σχέδιο διεθνούς ε, σύμβασης για τα πνευματικά δικαιώματα. Αν θα δίνονται στις βιβλιοθήκες όταν πρόκειται για ορφανά έργα. Στο που ετοίμασε η IFA. Εγώ βλέπω ένα πρόβλημα επίσης με την τροπολογία που αναφέρεται στο άρθρο 3 τροπολογία του εισηγητή και θέλω να ακούσω πώς ε, το εξηγεί ο εισηγητή. Τι εννοεί στο 75α όταν λέει ότι την ευθύνη την έχουν τα κράτη-μέλη. Στην τελευταία του τροπολογία, δηλαδή αριθμός 15 πρέπει να συζητήσουμε πολύ και με τους άλλους σκιώδες συζητητέ. Ειλικρινά είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή πάντως που μας ετοίμασε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, για τη σημαντική προσπάθεια. Ο κύριος Μάντερ θα αντιλάβει λάβει υπόψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Πρέντεργαστ. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσίαση τον κύριο Μάντερς θα πρέπει να προσέξουμε τη διάκριση στα αγγλικά ανάμεσα στη λέξη right holder και author, δηλαδή συγγραφέας και κάτοχος δικαιώματος. Και το θέμα ορισμού θα πρέπει να ρυθμιστεί σε επίπεδο κράτους μέλους, γιατί το άρθρο 3 τίνει να εννοήσει κάτι το οποίο... δεν είναι κατανοητό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 Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομος όσο ε, η προηγούμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ τον κύριο Μάντερς. Να πω ότι συμφωνώ μαζί του ότι το copyright είναι βασικό για να υπάρξει καινοτομία και ε, επένδυση σε μια εφάνταστη βιομηχανία, δημιουργική βιομηχανία και θα πρέπει να το αμύψουμε γιατί αλλιώς θα υπάρξει πραγματικά μείωση της δημιουργικότητας. Η καινοτομία είναι ζωτική για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες ψηφιακές πραγματικότητες, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην πρόσβαση στις αγορές και την αμοιβή των δημιουργών στο Ενωμένο Βασίλειο έχουν υπάρξει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σε κατηγορίες εις βάρος του Google για μονοπωλιακές ρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε εδώ και να υπάρξει η απαιτούμενη ισορροπία. Το ότι τα κράτη-μέλη έχουν την επιλογή εφαρμογής περαιτέρω μέτρων εφόσον το επιθυμούν είναι κάτι το οποίο εκτιμώ. Σαν παράδειγμα, η χρήση των ορφανών έργων για εμπορικούς λόγους μπορεί να επιτραπεί μόνο μετά από επιστάμενη έρευνα, όπως επίσης και η εθελοντική διεύρυνση αδειών χρήσης από συλλογικά όργανα. Ένας άλλος τομέας είναι η αμοιβή για τη χρήση των ορφανών έργων όταν βρεθεί ο ε, συγγραφέας. Η τροπολογία 15 ορίζει ότι όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν στο κράτος όπου έγινε η έρευνα. Ενώ να, θα πρέπει να μιλήσουμε για το κράτος μέλος το οποίο χρησιμοποιείται το έργο. Και ταυτόχρονα αν υπάρχει μία σύμβαση με άλλο σώμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το ορφανό αυτό σε εισαγωγικά έργο για μια άλλη χρονική περίοδο, αυτό γίνεται με μια νέα σύμβαση. Τώρα αυτό είναι λίγο τεχνικό. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Κύριε Άμστρομ, θέλετε να μιλήσετε για τους πρασίνους. Σας διορίζουμε θελοντή. Δεν διάβασα τη γνωμοδότησή του. Μου τη στείλατε, είπατε με mail, δεν μάλλον το χάσα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας αφορά και πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μιλάμε για εμπορικές χρήσεις, για μη εμπορικές συγγνώμη χρήσεις, δημόσια χρήση, βιβλιοθήκες κτλ. Εγώ θα ήλπιζα να είχαμε μία πρόταση για τα ορφανά έργα που να καθιστούσε ε, δυνατή την εμπορική χρήση, σαν παράδειγμα ένας ντοκιματαρίστας να μπορεί να χρησιμοποιήσει ιστορικά φιλμ, ιστορικές φωτογραφίες. Αυτή είναι μια εμπορική δραστηριότητα μεν, αλλά πολιτιστικά είναι ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα και οικονομικά θα μπορούσε να παρουσιάσει κάποιο ενδιαφέρον. Οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες θα πρέπει να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το πολυπίκυλο σώμα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, της πολιτιστικής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Δεν θα πω κάτι άλλο σχέση με αυτό. Να σχολιάσω αυτό που είπε ο κ. Μάντελ για τη βάση δεδομένων. Συμφωνώ μαζί του. Θα πρέπει οι τράπεζες δεδομένων να είναι εύκολα ανοιχνεύσιμες και λειτουργικές. Και το είπε και η κυρία Ρόιτοβα. Και η κυρία Ρόιτεβα λέει ότι δεν αναφέρεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χρηματοδότηση και όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσια μουσεία, με βιβλιοθήκες, είναι εξαιρετικά ιδρύματα όλα αυτά, αλλά δεν έχουν λεφτά και αν περι, κάποιος από εμά έχει, έχει την πρόθεση να περιμένει έτσι ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτά τα όργανα, δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί, γιατί εφόσον δεν επιτρέπονται εμπορικέ δραστηριότητες γύρω από αυτά τα έργα τα ορφανά, οι βιβλιοθήκες δεν έχουν και τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Το θέμα που έθεσε ο κύριος Φόξ για την εμπορική χρήση τίθεται εκ νέου. Ναι. Και όταν τερματίζεται μία σύμβαση και εμφανίζεται ξαφνικά ο κάτοχος του δικαιώματος, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί ακόμα και αν ψηφιοποιηθεί κάτι, και το χρησιμοποιήσουν εν μέρη αυτό το κάτι που θα ψηφιοποιηθεί, δεν παρουσιάζει ίσως την δυνατότητα που θα έπρεπε έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματικά εμπορική χρήση. Εν πάση περιπτώσει, ε, φοβάμαι ότι η έκθεση αυτή έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν μας αφορά. Um, any λοιπόν, κάποιο άλλο μέλος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και τους Σκιώδης για διάφορα χρήσιμα σχόλια. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φρόλιγκε για ένα μικρό σχόλιο και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Μάντερς να κλείσει τη συζήτηση. Uh, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενθαρρύνεται από την συζήτηση που είχατε εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας, όπως και από την χθεσινή συζήτηση που παρακολουθήσαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Αλλά και στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Υπάρχει γενική στήριξη στην πρόταση, αντιλαμβανόμαστε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται ότι συμμερίζεται τη δικιά μας ανάλυση, ότι πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε γρήγορα με το θέμα αυτό για να κλείσει το χάσμα, το κενό που υπάρχει και προκειμένου οι θησαυροί που έχουμε στα ευρωπαϊκά μας αρχεία, βιβλιοθήκες κτλ. να είναι διαθέσιμα στους ερευνητές μας, στους φοιτητές μας και στο στο γενικό κοινό. Όπως λέει και ο κύριος Μάντες, κάθε πρόταση της Επιτροπής επιδέχεται βελτίωση. Πράγματι, ακούσαμε ενδιαφέρουσες προτάσεις για βελτίωση σήμερα από τον εισηγητή σας και από τους κοιόδης εισηγητές. Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα. Θα τα εξετάσουμε πρώτα τα σχολιά σας και μετά μόνο πάνω σε μερικά θέματα που θυχτηκαν εδώ θέλω να σχολιάσω. Το πρώτο είναι αυτό που ακούσαμε από την κυρία Ρέτοβα και άλλους για το πεδίο εφαρμογή που περιορίζεται στα έντυπα έργα. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ε, από τα αρχεία και από Ινστιτούτο κιματογράφου πρέπει να βρεθεί κάποια λύση και για φωτογραφίες ατόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε δημοσιεύσεις, αλλά πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο περιπλέκει πολύ την πρόταση και ότι όντως θα σήμαινε καθυστέρηση στην νομοθετική διαδικασία. Συνεπώς, καλό θα ήταν να μην ζητήσουμε να επεκταθεί έτσι το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Έπειτα αναφερθήκατε στην εμπορική ή μη εμπορική χρήση. Φυσικά και θα μπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον να επιτραπεί και η εμπορική ή κάποιο είδου εμπορική χρήση. Τότε όμως χρειαζόμαστε μια διαφορετική πρόταση. Η καποιο ειδου εμπορικη χρηση τοτε όμω χρειαζομαστε μια διαφορετικη προταση η προταση μας είναι ξεκάθαρη. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να κάνουν την έρευνα και μετά να χρησιμοποιούν χωρίς να πληρώνουν και χωρίς να χρειάζεται να βάζουν στην πάντα χρήματα στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κάτοχος της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εμπορική χρήση, γιατί τότε εννοείται ότι ο κάτοχος ε, των πνευματικών δικαιωμάτων ε, τότε θα πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά που γίνεται εμπορική χρήση. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό εδώ να δούμε είναι ότι αυτό που επιτρέπει η οδηγία είναι την συνεργασία ιδιωτικού δημοσίου τομέα, δηλαδή μεταξύ βιβλιοθηκών και εμπορικών παραγόντων. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι οι βιβλιοθήκες δεν έχουν χρήματα και σήμερα μάλιστα που είμαστε σε οικονομική κρίση έχουν ακόμα λιγότερο από ό,τι είχα κατά το παρελθόν. Αλλά γι' αυτό και τους επιτρέπουμε, αφού έχουν κάνει την έρευνα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ορφανά έργα χωρίς πληρωμή. Και επιτρέπουμε επίσης τη συνεργασία τους με εμπορικούς ε, παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν ε, κατά τη διάρκεια αυτής της ε, ψηφιακής έκφρασης των έργων. Αυτό που κάνουν δηλαδή οι βιβλιοθήκες που περνάνε σε ψηφιακή μορφή τα ορφανά έργα. Δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει ανταγωνισμός του ιδιωτικού τομέα με τη βιβλιοθήκη η οποία φροντίζει για την ψηφιακή έκφραση. Κάτι άλλο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας, είναι το θέμα της βάσης δεδομένων. Και αυτό τέθηκε και πιστεύουμε ότι θα ήταν σημαντικό η έρευνα αυτή να γίνει απλή αλλά και νομικά ασφαλής. Αν έχουμε ένα δίκτυο βάσης δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα και να κοιτάξουμε και το θέμα των μεταφράσεων. Γιατί είναι αλήθεια ότι ένα όνομα μπορεί να είναι εντελώ διαφορετικό στη μία γλώσσα από ό,τι στην άλλη. Όπως επίσης και ο τίτλος ενός έργου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά μεταφρασμένος στις διάφορες γλώσσες. Οπότε η Επιτροπή πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη της και ίσως θα πρέπει να κάνουμε μία μελέτη σκοπιμότητας για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα τώρα. Αν ένας ε, συγγραφέας εμφανιστεί, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο θέλει να συνεχίσουν οι βιβλιοθήκες να χρησιμοποιούν το έργο του ή κατά πόσο θέλει, για οποιοδήποτε λόγο, να πάψει αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν ε, συχνά τέτοιες περιπτώσεις, όμως πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας και αυτές τις Αυτό που έχουμε στην πρότασή μας τώρα είναι, πιστεύουμε, η καλή λύση, αλλά σίγουρα επιδέχεται παρετέρω βελτιώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας και για την επικοδομητική προσέγγιση που έχετε απέναντι στην έκθεση. Ο κύριος Μάντας μήπως θέλει να κάνει μια σύνοψη και να μας πει και το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι. Συγγνώμη, ο κύριος Αμπάνσκι από την Πολωνική Προεδρία ήταν εδώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας ανέφερα πιο πριν. Έχουμε ένα πολύ καλό βιβλιαράκι εμείς εδώ με όλους τους εκπροσώπους της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Δεν ξέρω αν το έχετε όλοι. Μήπως θέλετε να πείτε και εσείς κάτι πριν κλείσουμε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Από το Συμβούλιο δύο λόγια. Συμφωνούμε ότι όντως υπάρχει μεγάλη ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα των ορφανών έργων. Πολλά από τα ζητήματα που ακούστηκαν έχουν συζητηθεί και στην σχετική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Οπότε πραγματικά συμμεριζόμαστε πολλές από τις απόψεις σας. Ε, προς το παρόν ε, προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε το συμβαστικό κείμενο της Προεδρίας ώστε να καλύψουμε κάποιες από αυτές τις ανησυχίες και συμφωνούμε με τον εισηγητή, τον κύριο Μάντερς, ότι η προστασία, η αποτελεσματική του, των πνευματικών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργική βιομηχανία. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν δημιουργούμε μηχανισμούς που επιτρέπουν τη χρήση ε, έργων χωρίς την έγκριση του κατόχου των αποβατικών δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες ε, ασφαλιστικές δικλείδες. Σίγουρα θα το μελετήσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπουμε στην υποβολή της ε, γνωμοδότησης από την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Εσύ είσαι αυτός που θα μας καθυστερήσει για να γιορτάσουμε τα γενέθλια της ε, συναδέλφου Βάιλερ με ένα ποτό. Οπότε να είσαι γρήγορος. Ε, η κυρία από την εκπρόσωπο τη Επιτροπή απάντησε πολλά από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Μόνο τη κυρία Ρόιτοβα έμεινε αναπάντητο για το σημείο 1-5α. Ίσως να πρέπει όντω να το αναδιτυπώσω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η ευθύνη για το κράτο μέλο είναι η νομική βάση, ότι δηλαδή ο χρήστη που χρησιμοποιεί το έργο από τη στιγμή που είναι γνωστό ο κάτοχος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ε, νομική βάση. Η ε, ερδελική έρευνα θα πρέπει να γίνει στο κράτο μέλο, αλλά ο χρήστη θα πρέπει να πληρώνει για τη χρήση του έργου. Εντάξει, θα το ανατυπώσω για να είναι πιο σαφέ. Για τα υπόλοιπα, Πρόεδρε, έχετε το χρονοδιάγραμμα. Εγώ έχω ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς. Ε, ελπίζω οι συνάδελφοι να κάνουν έτσι επικοδομητικές προτάσεις, να υποβάλουν τις ε, τροπολογίες τους. Άκουσα βέβαια τα σχόλια όλων, οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε λίγες εβδομάδες, θα είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάντερς. Λοιπόν, προθεσμία για τις τροπολογίες 26 Οκτωβρίου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα μελετήσουμε τις ε, τροπολογίες 21 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε θα υπάρξει ε, ψηφοφορία και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η, και η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει γρήγορα. Οπότε ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ και όλους για τα σχόλιά σας. Έχουμε και άλλο ένα σημείο στην εμμυρίστη διάταξη, αλλά έχω λάβει την ε, εκτελεστική απόφαση που λέει ότι θα σας, ε, και θα σας διανύμουμε ε, το κείμενο που αφορά την, ε, το σχετικό σημείο, οπότε θα μπορέσετε να το διαβάσετε με την άνεσή σας, γιατί υποσχέθηκα στην κυρία Βάιλερ ότι θα τελειώσουμε στην ώρα μας. Τελειώνουμε, κυρία Βάιλερ, τέσσερα λεπτά πιο νωρίς. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε στις 9 αύριο το πρωί και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη γνωμοδότηση για την εναρμόνιση της ιστορικής Αγορά. Ε, είναι από τα θέματα που ασχολείται η κυρία Φούλινγκ, οπότε μάλλον θα είναι μαζί μα και πάλι. Και έχουμε και ψηφοφορίε από τι 10 μέχρι τι 11. Μην ξεχάσετε τι κάρτε σα. Η κυρία Βάιλερ ήθελε να συναντηθούμε και μετά την συνεδρίαση. Μας έχει καλέσει όλους, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε κλείνουμε τη συνεδρίαση και θα τα πούμε έξω γιατί νομίζω ότι μας περιμένει ένα ποτό. Έξω από την αίθουσα. Οπότε, πέρα στις συνεδρίασεις και πάμε να πιούμε το ποτό.